Παρακαλώ, αποχωρήστε ησύχω για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Τώρα θα έχουμε την παρουσίαση του σχέδιου έκθεση για τον κανονισμό πλαίσιο με την κυρία Μπιόρκ, η συγγήτρια. Πρόκειται για ασφαλή άφηξη στις χώρες μας και για ανθρωπιστική εισδοχή και σχετικές πρωτοβουλίες, όπως επίσης και για την εμπειρία των χωρών μελών από τα διάφορα προγράμματα μετεγκατάστασης. Θα ζητήσω από την εισηγήτρια να μας παρουσιάσει το σχέδιο εκθεσής της. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Ησυχία για να ακούσουμε την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένω όντω να φύγει ο κόσμος. Πρώτα. Although if we keep pausing, people keep leaving slowly. That's the only thing. Let's start. Let's start. Ωραία, ας αρχίσουμε τότε. Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, τους ειδικού, τους ειδικούς επιτόπου και βέβαια και την γραμματεία της Επιτροπής μας ΛΥΜΠΕ που συνεργάστηκε μαζί μου και με την ομάδα μου. Όταν πρόκειται για το κοινό σύστημα σύλλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναθεωρούμε αυτή την εποχή, περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία. Τον καταμερισμό της ευθύνης πρώτα απ' όλα, Καλά, θα περιμένω μέχρι να υπάρξει περισσότερη ησυχία στην αίθουσα, λέει η συγγήτρια. Πρόεδρο, ξέρω ότι αυτά που συζητάτε είναι σημαντικά, αλλά έχουμε την εισηγήτρια η οποία μα παρουσιάζει την έκθεσή τη. Γι' αυτό σα παρακαλώ ησυχία. Ωραία. Θα επαναλάβω γιατί το πιο σημαντικό ήταν οι ευχαριστίες μου προς τους σκιώδεις εισηγητές και τη γραμματεία της ΛΥΜΠΕ που μας βοήθησαν. Το κοινό σύστημα σύλλου που αναθεωρούμε αυτή την ε, εποχή δεν ε, αναφέρει τίποτα για τη νόμιμη άφηξη μεταναστών και προσφύγων στις χώρες μας. Χρειάζονται λοιπόν ασφαλείς οδοί και γι' αυτό και ζητάμε νέες αποφάσεις από το Κοινοβούλιο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον ΟΗΕ, την ε, ε, Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ κλπ. Για να υπάρξουν όλο και περισσότερες ε, επανεκαταστάσεις και η επανεκατάσταση βέβαια θυμίζει λίγο αυτά που λέμε για την μετανάστευση, πρόκειται όμως για κάτι διαφορετικό, γιατί η επανεκατάσταση πρέπει να αναγνωριστεί σαν κάτι συμπληρωματικό. Δεν αντικαθιστά άλλες οδούς, είτε πρόκειται για ανθρωπιστικές θεωρήσεις βίζα, είτε πρόκειται για επανέναση οικογενειών κλπ. Η Επιτροπή του ΟΗΕ λοιπόν φτιάχτηκε στον ΟΗΕ μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακριβώς για να βοηθήσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έφυγαν από τα σπίτια τους εξαιτία του πολέμου. Υπάρχει σύμβαση της Γενέβης λοιπόν του 51, τα ξέρετε βέβαια, αλλά στην πρότασή μου έχω ένα πρώτο κομμάτι στο οποίο αναφέρομαι στην αρμοστή των ΗΠΑ για τους πρόσφυγες. Η πατερμοστή αυτή λοιπόν δημιουργήθηκε από τον ΟΗΕ προκειμένου να φροντίσει για την, για την επανεγκατάσταση που ήταν μία από τις λύσεις που βρέθηκαν τότε η επανεγκατάσταση προκύπτει όταν οι υπόλοιπες λύσεις έχουν ε, γίνει είτε η ένταξη στις χώρες υποδοχής μετά φτάνουμε στην επανεγκατάσταση. Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο προσφέρει προστασία και μία λύση διαρκείας για τους πρόσφυγες. Ο στόχος μου είναι διπλός. Αφενός να διατηρηθεί η ανθρωπιστική ιδέα της επανεκατάστασης και από την άλλη μεριά να ενισχυθούν οι προσπάθειες επανεκατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα χρειάζεται να αλλάξουμε κάπως τους στόχους, τις διαδικασίες, τις πρότασεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ξαναδούμε τις κατηγορίες στις οποίες έχουμε καταλήξει για την επανεκατάσταση. Η προτεραιότητα είναι να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο επανεκατάστασης. Όσον αφορά τους στόχους και τις διαδικασίες, νομίζω ότι πρέπει να βασιστούμε στις επιτυχείς περιπτώσεις επανεκατάστασης που είχαμε μέχρι τώρα και στις εμπειρίες των χωρών μελών. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος της ΥΠΑ Αρμοστίας ε, του ΟΗΕ είναι να συμμετέχει στις επανεγκαταστάσεις αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στο τι λειτουργεί καλά επί τόπου και να προβλέψουμε και για ρήτρες ασφαλείας στις διαδικασίες που εφαρμόζονται. Επιμένω στο γεγονό ότι η επανεκατάσταση είναι και ανθρωπιστικό μέσο για να βελτιωθεί η κατάσταση των προσφύγων. Ο ορισμός, η γλώσσα, θα δείτε, είναι πολύ πιο κοντά στην ύπατη αρμοστία για του πρόσφυγες του ΟΗΕ. Βέβαια, οι γεωγραφικές προτεραιότητες πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες για την επανεγκατάσταση, κάτι το οποίο το κάνει κάθε χρόνο ο Το κύριο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να αξιολογήσουμε πού χρειάζεται η επανεγκατάσταση είναι ακριβώς αυτό. Πρέπει να ενισχύσει τις προσπαθίες της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ερεσιμότητα τώρα για τη Συμφωνία Επανεστοχής και τον έλεγχο των ε, συνόρων συμπεριλαμβάνεται εδώ συγχρόνως με την στρατηγική σημασία της επανεγκατάστασης. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η επανεγκατάσταση και για άλλους σκοπούς για να ε, βρεθούν βιώσιμες λύσεις για περισσότερο κόσμο και για να ενισχυθεί η προστασία των προσφύγων. Όταν φτάνουμε στο θέμα της επιλογής, έχουν προσαρμοστεί, θα δείτε, προσαρμοζόμαστε με τις κατηγορίες της υπερσαρμοστίας του ΙΕ πολύ περισσότερο, έχουν τροποποιηθεί και τα κριτήρια αποκλεισμού για να ε, ανταποκριθούμε στο όσο προβλέπει η Σύμβαση της Γενέβης. Το πλαίσιο θα λειτουργήσει, ελπίζουμε, επιτόπου βάσει του διεθνούς δικαίου. Κριτήρια τώρα που λένε για κυρώσεις όσων παράνομα επερνούν τα σύνορα, κυρώσεις για πέντε χρόνια, πιστεύουμε εμείς ότι δεν ανταποκρίνονται. Ο ρόλος τώρα της τριμερής διαβούλευσης για την επανεγκατάσταση είναι μια συνάντηση αυτή όπου η ΥΠΑ και του με κυβερνητικέ οργανώσεις συναντιούνται κάθε χρόνο η Ανώτατη Επιτροπή για την Επεκατάσταση πρέπει να συμμετέχει ακριβώς εκεί και να συμμετέχει στις διεθνείς προσπάθειες προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει σημαντικά για να υπάρξει η επανεκατάσταση παγκοσμίω. Το πλαίσιο επανεκατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι διετέ και όχι μόνο ετέ, γιατί νομίζω ότι ο σχεδιασμό διευκολύνεται έτσι και για τι χώρε μέλη αλλά και για όλε. Κύριο στόχο μα με τη σύνταξη της έκθεσης αυτής είναι να ενισχύσουμε τις προσπάθειες επανεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια συγκεκριμένη πρόταση για νόμιμες οδούς, διότι η επανεγκατάσταση πρέπει να αυξηθεί. Τώρα που έχουμε και την κυβέρνηση Τραμπ μάλιστα, έχει γίνει το αντίθετο, έχει μειωθεί η επανεγκατάσταση. Πολλά μπορούν να γίνουν ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει το ρόλο της και την προσφορά της στην επανεγκατάσταση. Κάποιες χώρες μέλη είναι απρόθυμες να δημιουργήσουν νόμιμες οδούς εισόδου των προσφύγων. Και όλοι ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ακολουθούν μη ασφαλείς δρόμους με φοβερές απώλειες ζωής. Πράγμα από το οποίο αποφελούνται βέβαια πάνω από όλοι οι λαθροδιακινητές. Ένα τέτοιο πλαίσιο έχει νόημα εφόσον είναι αξιόπιστο. Όσον αφορά τα νούμερα, Συνεπώ, το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να φροντίσει τουλάχιστον 25% ετησίω να ανταποκρίνεται στις ανάγκες επανεκατάστασης με τον ΟΗΕ και τους άλλους εταίρους. 250.000 άνθρωποι δηλαδή μέσα στο 2017 και αυτό είναι κάτι που μπορεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ερχόμαστε τώρα στη συμμετοχή των χωρών μελών, η συμμετοχή τους παραμένει σε θελοντική βάση και στο δικό μου σχέδιο έκθεσης. Και αυτό για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με ένα σύστημα που λειτουργεί αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακροπρόθεσμα όμως, φυσικά, δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι δυνατόν στο κοινό σύστημα ασύλου να συμμετέχουν μερικώς μόνο μερικές χώρες να ε, δέχω τον έλεγχο στα σύνορα, αλλά να μην συμμετέχω στην επανεγκατάσταση. Επιπλέον, για τα εθνικά προγράμματα και τη σχέση τους με το ευρωπαϊκό. Το ζήτημα είναι να ενισχύσουμε κίνητρα για τις χώρες μέλη, ώστε να προχωρούν περισσότερο σε πράξεις επανεγκατάστασης. Πρέπει να τις ανθαρρύνουμε και να ενισχυθεί η συμμετοχή των χωρών μελών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πανεκατάστασης και χώρε που δεν έχουν εμπειρίες από επανεκατάσταση πρέπει να τι βοηθήσουμε με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, για παράδειγμα με άλλε χώρε μέλη, με τεχνική υλική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου που θα δημιουργηθεί. Και αν το ευρωπαϊκό πλαίσιο επανεκατάστασης αποθαρρύνει τις εθνικές προσπάθειες επανεγκατάστασης, δεν νομίζω ότι αυτό θα ήταν θετικό. Πάντως είμαι πεπισμένη ότι οι χώρες μέλη θα θελήσουν να βελτιώσουν την κατάσταση όσον αφορά τους πόρους και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επανεγκατάστασης. Και η επιτυχία του βέβαια θα κρυθεί από την αποτελεσματικότητά του και την ποιότητα. Χρειάζονται όπως είπα κίνητρα για τι χώρες μέλη προκειμένου να συμμετέχουν και η ισορροπία θα βρεθεί εφόσον οι χώρες μέλη έχουν 6.000 ευρώ, να τα κρατήσουν δηλαδή, που παίρνουν ε, πρόσφυγα από την ΑΜΙΘ, εφόσον συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επανεκατάστασης. Ένα άλλο ζήτημα που θα βρείτε στην έκθεσή μου είναι η βάση της ε, επανεκατάστασης αυτή καθεαυτή, γιατί θα το δείτε όταν πηγαίνετε και βρίσκετε τους ανθρώπους αυτούς και τους λέτε ορίστε θα σας μεταφέρουμε, τους φέρετε στην Ευρώπη και τους λέτε θα είσαστε ασφαλείς εκεί, έχετε την ευθύνη να δημιουργήσετε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον τους δώσετε και μια μόνιμη διαμονή. Και εδώ χρειάζεται να γίνονται περισσότερα από αυτά που τώρα διαπραγματευόμαστε. Προκειμένου όμως να το πετύχουμε, εγώ προτείνω οι χώρες μέλη να μπορούν να εκδώσουν τέτοιες ε, άδειες ε, παραμονής ε, μακροχρόνιες ή αόριστης διάρκειας. Να μπορούν να το κάνουν αυτό οι χώρες μέλη. Οπότε, επί της διαδικασίας. Έχω ζητήσει μια έκτακτη διαδικασία, ένα κατεπήγον. Είναι κάτι που ζητάει και η πατιαρμοστία του ΟΙΕ. Δεν το χρησιμοποιούν πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν πραγματικά χρειάζεται. Για τις δύο διαδικασίες τώρα που ήδη υπάρχουν, η τακτική και η έκτακτη, εγώ τις διατηρώ με κάποιες αλλαγές. Στην τακτική διευκρινίζω ότι υπάρχουν διαφορετικά στάδια επανεγκατάστασης. Γιατί πολλοί ρωτούν πώς θα λειτουργήσει αυτό. Οπότε έχουμε την ταυτοποίηση, την υποβολή των περιπτώσεων, την αξιολόγηση, την απόφαση και την καταχώρηση. Και όπως είπα και νωρίτερα, είναι ρόλος της είπα της ε, αρμοστίας του ΟΗΕ. Πρέπει όμως και το θέμα των ε, αδειών να είναι θέμα των χωρών μελών, να μπορούν ε, να τις δώσουν τις χώρες μέλη αυτό μετά την ε, άφηξη. Αν θέλουμε να δώσουμε μια θετική εικόνα της Ευρωπαϊκής Επανεγκατάστασης. Η αποθήκευση δεδομένων θα γίνεται αφού έχει ληφθεί θετική απόφαση. Κατά τα άλλα, στην υπόλοιπη διαδικασία δεν χρειάζεται τα δεδομένα να λαμβάνονται πριν αρχίσει η διαδικασία για να μην υπάρχει υπερβολικό γραφειοκρατικό βάρο για τις χώρες μέλη ή για την υπερτερμοστία του ΙΕ ή με τον τρόπο αυτό να δημιουργούμε υπερβολικέ προσδοκίες στους ετούντε. Οι χώρες μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το καθεστώ του προσφύγου εφόσον πιστεύουν ότι μέσα στα χρονικά όρια της διαδικασίας μπορούν να το κάνουν. Πρέπει να υπάρχει ευελιξία πάντως στη διαδικασία αυτή. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο για τις χώρες μέλη να μπορούν αν θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν, αλλά να μην είναι εξορισμού. Τέλος, οι εκτοπισμένοι. Ξέρω ότι πολλοί από εσά έχετε εκφράσει ανησυχίες από αυτού. Εγώ για τους εσωτερικά εκτοπισμένους το αναφέρω στην εκθεσή μου και λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι όλο και περισσότεροι. Και η διεθνή κοινότητα πρέπει να βρει δομέ και διαδικασίες για να στηρίξει και αυτούς που είναι εσωτερικά στη χώρα τους εκτοπισμένοι. Και ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε αυτό. Περιμένω τώρα και προσβλέπω στα σχόλια των συναδέρφων. Ευχαριστώ. Thank you very much, Madeline, for your work. Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σου σε αυτό. Τώρα θα ακούσουμε τους ε, σκιώδεις. Ε, όπου δεν υπάρχει σκιώδης ηγητής, ε, ίσως θα μπορούσε κάποιος άλλος συνάδελφος να τοποθετηθεί για να ακούσουμε τι έχουν να πούν όλες οι ομάδες. Ναι, ναι, σε βλέπω ότι είσαι εδώ. Ξέρω ότι το ΕΛΚ είναι εδώ. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Διασδαμέρα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη Μάλιν για το έργο της. Καταρχήν, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση η οποία προέρχεται από την Ισπανική καμπίνα, δεν έχει να κάνει με την Αγγλική καμπίνα. Από την Ισπανική καμπίνα συστηματικά και επανειλημμένα χρησιμοποιήθηκε ο όρος μετεγκατάσταση, δεν μιλάμε για μετεγκατάσταση, μιλάμε για επανεγκατάσταση. Και η διαφορά, και το λέω με παιδαγωγικούς όρους, είναι η εξής. Το να μεταγκαθαστήσω κάποιον είναι να τοποθετήσω αλληλέγγυα, ως εφημισμό το χρησιμοποιώ, όσους ε, ε, έχουμε να μεταφέρουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ η επανεγκατάσταση τι σημαίνει ότι δεχόμαστε και μοιράζουμε όσους είναι εκτός της Ένωσης. Αυτό είναι το αντικείμενο της έκθεσης της Μάλιν. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή τι κάνει, εγγυάται ένα σύστημα αφήξεων που είναι ανθρωπιστικό, αξιοπρεπές και μέσω σίγουρων οδών. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, θέλω να ευχαριστήσω την συγγήτρια για είναι πολύ ουσιαστικά σχολαστική δουλειά που κάνει. Θεωρώ ότι το ουσιαστικό για την Ένωση είναι να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα επαναγκατάστασης αποτελεσματικό, ρεαλιστικό και αλληλέγγυο πάνω απ' όλα. Και όπως ε, θα γνωρίζετε η Ευρώπη έχει το 23,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ σύμφωνα με τον ΟΣΑ. Και μόνο υποδεχόμαστε το 8% των προσφύγων του πλανήτη. Όπως γνωρίζετε, Πρόεδρε, εγώ και εσείς είχαμε το προνόμιο να μεταβούμε στον Καναδά και να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε το επιτυχές πρόγραμμα επανακατάστασης που έχουν εκεί, η διεισόμαση. Η χώρα αυτή, όπως ισχυρίζεται η Μάλη, στην έκθεσή της, δίνει ανδιαφυσβήτητη σημασία ε, στον ρόλο του ΟΗΕ. Στο ρόλο της ύπατης αρμοστίας. Και όπως θα έπρεπε να είναι και η δέσμευση και η χορηγία, αν θέλετε, της κοινωνίας των πολιτών και των ιδιωτικών φορέων σε ό,τι αφορά την επαναγκατάσταση. Σίγουρα αυτή είναι μία από τις ε, επτά πρωτοβουλίες ε, που ξεκίνησαν στα πλαίσια του νομοθετικού πλαισίου για την αναθεώρηση των συστημάτων ασύλου. Μάλιν, έχω σκεφτεί πάρα πολύ το θέμα της ε, κατεπίγουσας ε, διαδικασίας και εγώ νομίζω ότι όπως και εσύ είναι γελίο να θεωρήσουμε ότι οι τέσσερις μήνες ε, είναι μια περίοδο κατεπίγουσα. Αν περιμένουμε τέσσερις μήνες θα γίνει κάτι θανατηφόρο. Έτσι λοιπόν, εγώ δεν θεωρώ ότι το κατεπήγον είναι τέσσερι μήνε. Ταυτόχρονα λαμβάνω υπόψη την ε, ισορροπία που προσπάθησε να βρει η συγγήτρια για να δώσει κίνητα, κίνητρα στα κράτη-μέλη και να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα επαναγκατάστασης της Ένωσης, όπως και τα εθνικά προγράμματα για τη χώρα μου, είναι θεμελιώδες και το εθνικό πρόγραμμα, γιατί έχουμε ισπανόφωνους αδελφούς που υποφέρουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μάλιν, θα καταθέσω 8 είναι επικοδομητικές τροπολογίες και μπορείς ε, να βασιστείς πάνω μου για πλήρη συνεργασία. Ευχαριστούμε κύριε Δίας Δεμέρα και σας ευχαριστούμε που μας αποσαφηνίσατε ουσιαστικά και τους δύο όρους, επανεγκατάσταση και μετεγκατάσταση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σας ευχαριστούμε που θέσατε και το θέμα της ε, αντιπροσωπείας στον Καναδά. Αν μπορούμε να προωθήσουμε κάποια από τα μοντέλα που είδαμε, στα πλαίσια αυτής της αποστολής, ε, σίγουρα θα ήταν καλό γιατί ήταν προοδευτικά αυτά τα μοντέλα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω γιατί έχουμε μόνο 45 λεπτά. Ζητώ συγγνώμη, όμως ε, θα εγγυηθώ ότι όλοι θα μιλήσουν. Δεν είναι εδώ και τυπέρι από τους σοσιαλιστές. Κάποιος άλλος μήπως θέλει το λόγο. Μήπως ε, θέλετε να πάρετε το χρόνο για τους σκιώδε, ή Μπριγκίτ και ο Φερνάντο, όποιος ε, θέλει. Εγώ θα πω μια λέξη μόνο και ο Χουάν μπορεί να προσθέσει κάτι. Θα ήθελα να πω ότι εκπλήσωμαι κάπως που χρειάζεται να μιλήσουμε για επανεγκατάσταση. Αν θέλετε να ζητήσετε, αν θέλει κάποιος να ζητήσει προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προέρχεται από μια χώρα με την οποία δεν έχουμε συμφωνία απαλλαγής θεώρησης, η μόνη δυνατότητα κάποιου είναι να φτάσει παράνομα που δεν είναι έγκλημα, ακόμη και αν ε, κάποιοι το πιστεύουν. Έτσι λοιπόν, αν ε, θέλεις ε, να είσαι σίγουρος για το ποιος έρχεται και θες να βοηθήσεις τους ανθρώπους να γλιτώσουν από τα βασανιστήρια και τον πόλεμο και τις διώξεις, η μόνη δυνατότητα είναι να οργανώσεις επαναγκατάσταση. Έτσι λοιπόν, αν είναι όλα τα θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά ζητούν άσυλο και χρειάζονται πράγματι προστασία, γιατί αν εργαζόμαστε με την επαναγκατάσταση δεν θα σταματήσει εντελώς σε καμία περίπτωση τους ανθρώπους που προσπαθούν να διαφύγουν από δύσκολες συνθήκες στη χώρα τους αλλά θα ελαχιστοποιήσει τις δυσκολίες και ε, ουσιαστικά θα καταφέρει και ένα κτύπημα ε, στους διακινητές. Εγώ βέβαια δεν είμαι τόσο αισιόδοξη αλλά πραγματικά πιστεύω τα κράτη-μέλη θα συνειδητοποιήσουν ότι ότι αυτό είναι ένα πολύ καλός τρόπος να αναλάβουμε την ανθρωπιστική μας ευθύνη και να δώσουμε προστασία στους ανθρώπους που προσπαθούν να γλιτώσουν τον πόλεμο, την πολιτική δίωξη και τα βασανιστήρια και να έχουμε και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες ότι οι άνθρωποι που έρχονται είναι πραγματικοί πρόσφυγες που ζητούν προστασία. Έτσι λοιπόν, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω οποιοδήποτε επιχείρημα από τα κράτη-μέλη που αντιστέκονται στην ιδέα αυτή και επειδή πάντοτε αυτό είναι το πρόβλημα σε όλες τις συζητήσεις, η επαναγκατάσταση δεν είναι η μόνη λύση. Βεβαίως θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα εμφανίζονται στα σύνορά μας και θα πρέπει να εργαστούμε και σε σχέση με την άσχημη κατάσταση που επικρατεί σε κάποιες από τις τρίτες χώρες. Η επαναγκατάσταση λοιπόν είναι ένα σημαντικό στοιχείο του πακέτου ασύλου και ελπίζω τα κράτη-μέλη να εργαστούν σε αυτό. Ευχαριστώ. Ε, τώρα κάτι. Ε, έδωσα το λόγο σε ε, δύο συναδέλφους του S&D για να δούμε λοιπόν την άποψη, την δεύτερη άποψη. θα είμαι σύντομος. My way out to the θα είμαι σύντομος. τυχαία συζητήσαμε και αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας. θα ήθελα περίμενα τους σκιώδεις ε, να ε, συζητήσουν για αυτό. Ε, όμως ε, δεν υπάρχουν ισχυώδεις που θα θέλουν να κάνουν σχόλιο, όμως από πλευράς μας θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι θα έχουμε πλήρη συνεργασία πάνω σε αυτό. Δεν είμαι ε, σκιώδης σε αυτή την αναφορά, στη συγκεκριμένη αναφορά, όμως είμαι ε, γνωμοδότης στην αναφορά και τις θεωρήσεις έτσι λοιπόν, ασχέτως των τεχνικών των τεχνικών λεπτομεριών ε, και τη βελτίωση του ζητήματος ε, στι ε, τροπολογίε θα πρέπει να είμαστε και πολιτικοί. Θα πρέπει πολιτικά να αντιμετωπίσουμε και την, και την άλλη πλευρά τη συζήτηση που είναι το Συμβούλιο. Για ποιο λόγο εξετάζουμε την μεταγκατάσταση και την επενεγκατάσταση, για ποιο λόγο εξετάζουμε εκ νέου τα όσα αποφασίστηκαν στην προηγούμενη θητεία, απλούστατα διότι το Συμβούλιο τα κράτη-μέλη συγκεκριμένα, κυβερνήσεις αυτών δεν τηρούν την νομοθεσία. Η επανεγκατάσταση δεν έχει εφαρμοστεί. Έχουν υπάρξει προγράμματα και αποφάσεις οι οποίες δεν εφαρμόζονται και για αυτόν τον λόγο επανεξετάσουμε όλο αυτό το ζήτημα διότι η επανεγκατάσταση δεν λειτουργεί ούτε και η μετεκατάσταση και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να κινηθούμε πολιτικά πάνω σε αυτό το ζήτημα. Επιπλέον, το να δημιουργήσουμε μια θέση ε, του Κοινοβουλίου θα πρέπει στρατηγικά να προχωρήσουμε προς τα εμπρός όταν το ζήτημα αφορά την, ε, τον τριμερή διάλογο ε, που είναι η τελευταία διαδικασία που αφορά την, ε, την υιοθεσία της συγκεκριμένη νομοθεσίας. Η νομοθεσία θα πρέπει να τηρηθεί από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ και τώρα περνάμε στην κυρία Helga Stevens. Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε ναι, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει ως τώρα. Βλέπω ότι υπάρχουν συνολικά 125 τροπολογίες, δεν είχα το χρόνο να τις διαβάσω όλες ε, και αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο ε, να δηλώσω κάτι διότι δεν τις διάβασα όλες. Αδειμονώ όμως να υπάρξει ένας επικοδομητικός και επικοδομητικός ε, διάλογος ε, στις συναντήσεις με τους ε, σκιώδεις και πιστεύω ότι η πρόταση δεν θα αλλάχθεί πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά χρειάζονται κάποιες μικρές αλλαγές. Σε βασικό επίπεδο όμως νομίζω ότι η πρόταση είναι μια χαρά, όμως θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί εν συνεχεία. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να αποφύγουμε ε, το να διπλασιάσουμε το έργο που έχουμε να κάνουμε με την ύπατη αρμοστία. Ε, θα πρέπει να κάνουμε τη βέλτιστη χρήση των πόρων που έχουμε Επιπλέον θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να ε, τεθεί ένα ανώτατο όριο ε, στους, στον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να ε, επανεγκατασταθούν στο χρονικό διάστημα που έχουμε. Είναι μια διαφορετική συζήτηση, όμως είναι σημαντική που πρέπει να κάνουμε για να διατηρήσουμε την υποστήριξη των πολιτών στην επανεγκατάσταση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους. Ευχαριστώ πολύ. Και η Σεσίλια Γουρξομ για το Άλντε. Ευχαριστώ πολύ εκπροσωπώ ε, την ε, Ρουή Μισελ που είναι σκιώδης και γι' αυτό το λόγο θα μιλήσω γαλλικά. Ο κύριος Μισελ λοιπόν ευχαριστεί πολύ την εισηγήτρια για το σχέδιο εκθεσής της όπως επίσης και για τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους σκιώδης εισηγητές. Η ανταλλαγή αυτή καταδεικνύει ότι υπάρχει πραγματική βόληση ώστε να προσφέρουμε μια πρόσθετη αξία στον προτινόμενο κανονισμό. Η επανεκατάσταση είναι ένα μέρος της λύσης που μπορεί να προσφέρει στην προσφυγική κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Λουί Μισελ λοιπόν έχει εμπιστοσύνη, είναι πεπισμένος ότι θα είμαστε επικοδομητικοί και φιλόδοξοι στην εκπόνηση μηχανισμών βάσει των οποίων ο καθένας πρέπει να αναλάβει το δικό του μερίδιο ευθύνης και εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της Μόλιν Μπιόρκ και των άλλων σχεδόν εισηγητών προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα είναι στο ύψος αυτών που ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από την αρχή της μεταναστευτικής κρίσης, δηλαδή την εκπόνηση και την ενίσχυση νόμιμων οδών για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι χρειάζονται διεθνή προστασία. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ωραία. Θα είναι πολύ περήφανος, Σεσίλια, για σας ο Λουί Μισελ. Ωραία. Εκ μέρους των Πρασίνων. Σάλβιο, θα μιλήσετε εκ μέρους των Πρασίνων. Δεν έχουμε η κυρία Σαγκετίνη είναι κανονικά για τους πράσινους, αλλά δεν είναι εδώ. Κανείς από το EFTD. Ωραία. Τότε, οι ευρωβουλευτές που θέλουν το λόγο, η κυρία Αλμπιόλ πρώτα. Α, υπάρχει σκιώδης από τους πράσινους. Συγγνώμη, δεν σας είχα δει. Αλλάξατε πάλι τα μαλλιά σας. Γι' αυτό δεν σας γνώρισα, ξυριστήκατε. Λυπάμαι, γι' αυτό δεν σας γνώρισα. Ήρθατε εγκόγνητο. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, είμαι τροπαλός, γι' αυτό δεν θέλω να με γνωρίζουν, γι' αυτό αλλάζω στυλ κάθε τόσο, λέει ο κύριος Φεράρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια. Ας κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις και εμείς από την δική μα ομάδα. Η επανακατάσταση θα πρέπει να γίνει ανθρωπιστικό εργαλείο και όχι διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ουσιαστικά καταδικάζουμε την ε, σύνδεση μεταξύ ε, των ανθρώπων προς επανακατάσταση και των ε, δικτών τη καταμέτρηση των μεταναστών. Έτσι λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να συνδέσουμε το θέμα με την διαχείριση των μεταναστευτικών στι τρίτε χώρε Κατά την άποψή μα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντλήσει τα περισσότερα διδάγματα και συμφωνούμε στο να καταργήσουμε κάθε αναφορά στη συμφωνία με την Τουρκία ως μοντέλο προς ακολούθηση βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια έκτακτη διαδικασία επανακατάστασης προς προτείνεται και αυτό να μπορέσει να βοηθήσει όσους βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Εμείς θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι σε σχέση με τον αριθμό ατόπων προς επανεγκατάσταση σε και το ότι πρέπει να συνεισφέρει η Ένωση στις παγκοσμίες ε, ανάγκες. Μόνο συγκεκριμένοι στόχοι μπορεί να κάνουν συγκεκριμένο αυτό το εργαλείο και πρέπει να συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία, κάτι που έλειπε μέχρι τώρα και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχει και ο αρμόδιος οργανισμός ε, ε, ένα κατάλληλο ρόλο για την επανεκατάσταση και επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να υπάρχει και παρουσία του οργανισμού στις τρίτες χώρες έτσι ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία. Τέλος, ε, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε την επαναγκατάσταση με άλλα εργαλεία όπως η οικογενειακή επανένωση. Εδώ συμφωνούμε με την συγκήτρια με την αναγκαιότητα να χρησιμοποιούμε την επαναγκατάσταση για να γίνεται η οικογενειακή επανένωση μόνο όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Κατά τα λοιπά, Είμαι στη διάθεσή σας για να βοηθήσω για να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, οι ευρωβουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο ατομικά, μεμονωμένα, παρακαλώ κυρία Βιόλ, επιτέλους σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επανεγκατάστασης αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της νέας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το άσυλο. Είναι μια πρόταση που βασίζεται στο ότι θα πληρώνουν τρίτες χώρες για να φυλάνε εκείνες τα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά η εγκατάσταση γίνεται σαν μία ρήτρα, σαν μία σύμβαση, όπου εμείς πληρώνουμε και κάποιοι άλλοι ελέγχουν τα δικά μας σύνορα. Παίρνουν ε, ανθρώπους, φέρνουν, ε, ε, φυλακίζουν τους παράνομους. Τελικά είναι εκείνοι που αναλαμβάνουν τη δικιά μας πολιτική ασύλου. Σύμφωνα με την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής λοιπόν, η πανεγκατάσταση δεν είναι ανθρωπιστικό μέσο εκτακτής ανάγκης αλλά αποτελεί ένα εργαλείο ελέγχου της μετανάστευσης μέσω συμφωνιών με τρίτες χώρες για να ε, διώχνουμε πιο εύκολα από τις δικές μας χώρες τους μετανάστες. Έτσι λοιπόν εμείς είμαστε επικριτικοί ε, στην πρόταση αυτή της Επιτροπής. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Γιώργο για την δικιά της πρόταση. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τελικά δεν επιτρέπει την επανεγκατάσταση σε ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν παράνομα τα τελευταία πέντε χρόνια να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια πρόταση που για μας αντιβαίνει στη Σύμβαση της Γενέβης η έκθεση της κυρίας Μπιόρκ υπογραμμίζει τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της επανεκατάστασης που δεν μπορεί να αντικαταστήσει άλλους τρόπους άφηξης μέσω νόμιμων οδών όπως ζητούμε και η έκθεση πηγαίνει στη γραμμή που λέει ότι οι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Είναι έκθεση που ξεκαθαρίζει ότι η επανεγκατάσταση δεν μπορεί να εξαρτάται από μεταναστευτικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να προσφέρει στους ανθρώπους αυτούς που επανεγκαθιστούνται στις χώρες μας μόνιμη άδεια παραμονής. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Μπιόρκο για το έργο της στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, ο κύριος Ράντε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα μόνιμο σύστημα επανεκατάστασης μεταναστευτών που να συνοδεύεται από κέντρα επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου στις χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί καταβλισμούς προσφύγων σε άλλες χώρες και τις βοηθάει όπως βοηθάει και οποιαδήποτε χώρα υποδέχεται πρόσφυγες από τη Συρία και αλλού. Γι' αυτό λέω ότι δίπλα στους καταβλισμούς αυτούς πρέπει να υπάρχουν κέντρα όπου όσοι θέλουν να αποκτήσουν το καθεστώς του πρόσφυγα να, του, να μπορούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου βάσει του ΟΗΕ και τα λοιπά. Και αν υπάρξει θετική απόφαση στην αίτησή τους αυτή για άσυλο, να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει δηλαδή να προσέχουμε μόνο τις χώρες που βρίσκονται στα δικά μας εξωτερικά σύνορα. Έτσι θα μπορέσουμε να σώσουμε εκατοντάδες ζωές, γιατί οι άνθρωποι αυτοί θέλουν διεθνή προστασία και δεν θα δοκιμάζουν να διασχίσουν τη Μεσόγειο με επικίνδυνου τρόπου, αλλά με ασφάλεια εφόσον έχουν υποβάλει την αίτηση ασύλου του με ασφάλεια στι χώρε όπου βρίσκονται. Έτσι εμείς θα μπορούμε να ελέγξουμε και για την ασφάλεια τα άτομα αυτά πολύ πριν μπουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι και οι Ευρωπαίοι πολίτες θα νιώσουν ότι είναι περισσότερο ασφαλείς. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι το μόνιμο σύστημα επανεγκατάστασης θα προσφέρει πολλά ε, στους ετούντες άσυλο, πολύ περισσότερα από όσα τους προσφέρουν τώρα οι χώρες μέλη. Συγχρόνως βέβαια είναι δύσκολο να δεχτώ την πρόταση της εισηγήτριας που λέει ότι οι χώρες μέλη μπορούν να αποκλείσουν από το σύστημα άτομα τα οποία θεωρούν ότι απειλούν την ασφαλειά τους. Είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο, ενώ λέμε ότι θα μπορούν άλλοι από τρίτες χώρες να μπορούν να έχουν μόνιμη άδεια παραμονής. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ο κύριος Ντεπρέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα δεν θέλω να πω γενικότητες. Συμφωνώ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με την εισηγήτρια. Και συμφωνώ και με τα όσα τόσο καλά είπε στα γαλλικά η συνάδελφος ο Σεσίλια Βελστρόμ που μετέφερε τις παρατηρήσεις του κ. Λουί Μισελ. Τώρα, εγώ έχω μια παρατήρηση και μια ερώτηση. Πρώτον, είμαι σκιώδης για τον προπολογισμό όσον αφορά ακριβώς αυτό το ζήτημα της επανεκατάστασης. Και προσωπικά δυσκολεύομαι με την πρόταση με την οποία φαίνεται να συμφωνούν οι ομάδες που λέει ότι για τα εθνικά προγράμματα θα συνεχίζαμε να δίνουμε 6.000 ευρώ στις χώρες αυτές ανά άτομο το οποίο αναλαμβάνουν για διεθνή προστασία στις χώρες τους, ενώ θα υπάρχουν 10.000 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Κοιτάξτε, Πρόεδρε, υπάρχει ένα θέμα αρχής εδώ. Συμφωνώ οι ευρωπαϊκές επιστώσεις να βοηθούν στη χρηματοδότηση δράσεων που γίνονται στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Δεν βλέπω όμως για ποιο λόγο ευρωπαϊκές πιστώσεις να βοηθούν οικονομικά για να στηρίξουν μια πολιτική που εντελώς αυτόνομα εφαρμόζουν κάποιες χώρες μέλη, ακόμα και αν είναι μια απόλυτα καλή και θεμητή πολιτική αυτή. Ε, πρόκειται για τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν πρέπει να περιορίζεται σε δράσεις που αποφασίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή που τέλος πάντων εντάσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια ερώτηση από την οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Οι χώρες μέλη μπορούν να αποφασίζουν ό,τι θέλουν, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι πρέπει να είναι συνεπές με τον εαυτό του. Τώρα, για το θέμα της θεώρησης είμαι σιώδης εισηγητής και έχω μια ερώτηση. Προβλέπετε για το σύνολο όσων θα ενταχθούν στην επανεγκατάσταση να έχουν ένα έγγραφο στα χέρια τους ευρωπαϊκό το οποίο σε όλες τις χώρες ή το αφήνουμε αυτό στην εκτίμηση της κάθε χώρας μέλος να αποφασίσει τι είδου ταυτότητα θα δώσει στους ανθρώπους αυτούς για να μπορούν να κυκλοφορούν τη διάρκεια θα έχει το έγγραφο αυτό, για παράδειγμα. Εγώ νομίζω ότι αν πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πρέπει και οικονομική αρρωγή να είναι ευρωπαϊκή αντίστοιχη, αλλά και η ταυτότητα που θα παίρνουν τα άτομα αυτά να δείχνει ότι πρόκειται για πρόγραμμα ευρωπαϊκού χαρακτήρα αυτό στο οποίο συμμετέχουν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλό είναι να τα ακούμε τώρα σε αυτό το στάδιο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που αναφερθήκατε και στα δημοσιονομικά. Και για πριν να ξαναδώσω το λόγο στη Μάλιν. Έχουμε τον κύριο Λενάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Εγώ εξεπλάγει ότι μόνο τα 14 από τα 28 κράτη-μέλη έχουν προγράμματα επέμβαση που λειτουργούν. Όμω, νομίζω ότι η ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάσταση όντω υπάρχει. Σε σχέση με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία εκεί. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για το έργο της. Ε, Απλά ήθελα να ξέρω πόσο εφικτά είναι όλα αυτά. Είδαμε ότι η επαναγκατάσταση έχει κάπως ε, ξαναρχίσει, αλλά ενθουσιασμός στα κράτη-μέλη δεν είναι πολύ υψηλός. Υπάρχει ένα δύσκολο ζήτημα για το αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικού ή εκούσιο χαρακτήρα. Η συγγήτρια διάλεξε τον εκούσιο χαρακτήρα, όμως ε, ταυτόχρονα έχει θέσει το στόχο των 250.000. Ε, δεν ξέρω λοιπόν αν ένας εκούσιος χαρακτήρας ε, συνάδει με το στόχο των 250.000, αν θα είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Εδώ προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε και εφικτά αποτελέσματα. Επίσης, πώς η οικογενειακή επανένωση εντάσσεται σε αυτό το πρόγραμμα επανακατάσταση στην Ολλανδία το 2016. Είχαμε περίπου 30.000 αιτήματα σύλλου και 30.000 άνθρωποι ήρθαν με, δια οδού μέσω της οικογενειακής επανένωσης ε, έφτασαν στην Ολλανδία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προθέσουμε και αυτές τις νομικές οδούς. Το κείμενο επίσης συγκρίνει την επανακατάσταση με το 2015. Υπάρχει, υπήρχαν τότε ένα εκατομμύριο άτομα που μπήκαν παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορώ να φανταστώ ότι ακόμη και αν δεν, είναι, δεν φαίνεται καλά κράτη-μέλη που είχαν μεγάλες εισρωές ε, προσφύγων, ε, ε, να, δεν, να επενδύουν ε, πάρα πολύ σε πολιτική επαναγκατάσταση. Ε, βλέπουμε ότι από τη μία έχουμε αυτή την πολιτική και από την άλλη συμφωνίες ε, για την παράτυπη μετανάστευση. Νομίζω ότι όλα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται εδώ. Και τέλος, Βάσει του ΑΕΠ μας κάνουμε έναν υπολογισμό. Όταν ε, μιλάμε για τους μηχανισμούς μεταγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνουμε το ΑΕΠ 50% και τον πληθυσμό άλλο 50%. Έτσι λοιπόν, ίσως αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσουμε και το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε όχι μόνο μια ευρωπαϊκή, αλλά μια παγκόσμια προσπάθεια. Γιατί αν όλα όσο προτείνουμε εδώ λειτουργήσουν, πάλι θα μιλάμε μόνο για το 25% ε, των ανθρώπων που έχουν προσδιοριστεί ως πρόσφυγες από την UNHCR, από την υπατερμοστία. Θα πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι έχουν ε, προσδιοριστεί για επανακατάσταση από την υπατερμοστία θα βρουν μια θέση. Ευχαριστώ. Είμαστε κάπω ε, πιεσμένοι από τον χρόνο και κατόπιν έχουμε και την έκθεση για τον μηχανισμό του Δουβλίνου. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο τη Κομισιόν πριν εξάδωσε το λόγο στην εισηγήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια, ευχαριστώ και τους βουλευτές. Να πω δύο λόγια και από την Κομισιόν. Η Κομισιόν ε, εκτιμά τη συνολική υποστήριξη για ε, το πλαίσιο επανεγκατάστασης και τη συμφωνία επί των ιδίων στόχων που θα πρέπει να προωθήσει το πλαίσιο αυτό. Απλώς να αναφέρω ότι μεταξύ άλλων στοιχείων που έχουμε στην επανεγκατάσταση. Η πρόθεση βασίζεται στα σημερινά συστήματα επανεγκατάστασης, τα οποία ε, λειτουργούν, δρομολογούνται, θα δείτε ότι πάνω από τα δύο τρίτα των ε, συμπεφωνηθέντων αριθμών έχουν ήδη επαναγκατασταθεί. Έχουμε περίπου 15.500 ανθρώπους που έχουν επαναγκατασταθεί από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Κάποια στοιχεία να αναφέρω σε σχέση και με τόσο όσο η Κομισιόν συμφωνεί πλήρω ότι ο ρόλο τη υπερτισερμοστία ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, γιατί είναι κεντρικό εταίρο στην επανεγκατάσταση. Έτσι λοιπόν θέλουμε να εργαστούμε περαιτέρω για να το διευκρινίσουμε αυτό στο ίδιο το κείμενο, για να διασφαλίσουμε ότι είναι σαφέ, ότι είναι απαραίτητο εταίρο ε, η υπερδεσμοστία. Η επανεγκατάσταση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προσφορά διεθνούς προστασίας, την παροχή διεθνούς προστασίας, είναι αυτός ο υπαριθμόν ένα στόχος. Όμως η Κομισιόν πιστεύει ότι η επαναγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στρατηγικά για να ενθαρρύνουμε τις τρίτες χώρες να αυξήσουν την ικανότητά τους για την υποδοχή και την παροχή προστασίας, έτσι ώστε να αυξήσουμε και την παγκόσμιο μερισμό ευθύνης δυνάμει της δήλωσης της Νέας Υόρκης. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η επαναγκατάσταση μπορεί να είναι ένα εργαλείο για καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης ε, σύμφωνα με το άρθρο 4 της πρότασής μας. Ορισμένα στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να θεωρηθούν ως παράγοντες ε, όταν θα αποφασίζουμε επί χωρών και περιοχών όπου θα λάβει χώρα η επαναγκατάσταση. Η επαναγκατάσταση λοιπόν είναι σημαντικό εργαλείο για την επιτεύξη διεθνούς προστασίας, όμως δεν ε, υπάρχει ε, σωστικό δικαίωμα για κάποιο άτομο για επαναγκατάσταση. Γι' αυτό η επαναγκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει κάποιον ευρύτερα στοιχεία μη επιλεξιμότητας σε σχέση με αυτά που έχουμε στη συνθήκη της Γενέβης. Όταν μιλάμε για αποκλεισμό στην πρόταση, δεν μιλάμε για αποκλεισμό από τη χορήγηση διεθνούς προστασίας, αλλά για αποκλεισμό ή αν θέλετε μη επιλεξιμότητα για την επαναγκατάσταση. Παραδείγματο χάρη, δεδομένη τη φύση τη επαναγκατάσταση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποκλείσουν από την επαναγκατάσταση άτομα για τα οποία έχει ε, εκδοθεί ε, ουσιαστικά καταχώρηση, στο, έχει υπάρξει καταχώρηση στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν ή αν είναι αντικείμενο άρνησης εισόδου τα άτομα αυτά. Η Κομισιόν συμφωνεί ότι το πλαίσιο θα πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της διακήρυξης της Νέας Υόρκης, να αυξηθούν οι νόμοι μεσοδοί και μέσω της επαναγκατάστασης Πιστεύουμε όμως ότι δεν θα ωφελήσει να έχουμε μια δεσμευτική κλίμακα επαναγκατάσταση στο πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια. Αντίθετα, προτείνουμε ένας μέγιστος ενότητας αριθμός να συμφωνηθεί, ετησίως να συμφωνείτε βάσει συζητήσεων μεταξύ των ε, κύριων εταίρων στη διαδικασία και φυσικά και του Κοινοβουλίου. Για τον προπολογισμό, η Κομισιόν ε, συμφωνεί απόλυτα με το σχέδιο γνωμοδότηση τη Επιτροπή Προπολογισμών. Θα πρέπει να έχουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο, πρέπει να έχουμε επαρκεί πόρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη για την επαναγκατάσταση. Αυτό απαιτεί στο να διατηρήσουμε τους περιορισμένους πόρους ε, που έχουμε στη διαθεσή μας. Ο προπολογισμό λοιπόν της Ένωσης θα πρέπει να υποστηρίζει την επαναγκαταστήση μέσω καταποκοπή ποσών ε, που ε, δίνονται σύμφωνα με κοινά κριτήρια επιλεξιμότητας ή αποκλεισμού και θα συμφωνούνται υπό κοινέ δομές που προβλέπει το πλαίσιο. Υπάρχει, υπάρχουν κάποια κονδύλια για την επανακατάσταση και υποτεθνικά προγράμματα, όμως αυτά είναι πέρα από τα καταποκοπήν ποσά. Μέσω των εθνικών προγραμμάτων μπορούμε να υποστηρίξουμε τεχνικά προγράμματα δίνοντας κονδύλια στα κράτη-μέλη για να δημιουργήσουν υποδομέ για να βοηθήσουν την επανακατάσταση. Όταν μιλάμε για καταποκοπήν ποσά, μιλάμε για τη σύνδεση μεταξύ του ευρωπαϊκού προπολογισμού και του ευρωπαϊκού πλαισίου. Και τέλο, η συνέπεια με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Στην πρότασή μας έχουμε το ίδιο καθεστώς για τους ανθρώπους ε, που επανεγκαθίσταται. Αυτό προβλέπεται και για άλλους ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίες. γιατί μιλάμε για τις ίδιες ανάγκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και να δώσουμε πάλι το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για όλες ε, τις συνεισφορές. Καταρχήν ε, θέλω να πω ότι συμπεραίνω ότι υπάρχει πολλή υποστήριξη για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επαναγκατάστασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προς αυτό κατευθυνόμαστε. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι θέλουμε ασφαλείς οικονομικές οδούς για την Ευρώπη, το νοούμε. Σε, προς, εκεί, προς αυτή την κατευθύνση θα εργαστούμε εδώ σε αυτό τον οίκο. Και επανειλημμένως το έχουμε πει. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε προς αυτό. Σημειώνω λοιπόν ότι υπάρχει πολλή υποστήριξη σε αυτή την προσέγγιση. Σημείωσα όλα τα διάφορα σχόλιά σας και τις ανησυχίες σας. Θέλω να κάνω όμως ένα γρήγορο σχόλιο για κάποια θέματα που αναφέρθηκαν και από τον συνάδελφο στην Επιτροπή Προεπιλογισμών. Και εγώ το είχα σκεφτεί φυσικά και το είχαμε συζητήσει και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών. Νομίζω ότι ειδικά τώρα όταν μιλάμε για φιλοξενία προσφύγων πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ξέρουμε ότι δεν είναι οι 6-10 που θα καλύψει το κόστος, θα καλύψει το κόστος ε, της υποδοχής προσφύγων. Αλλά το να αφαιρέσουμε συμβολικά αυτό το ποσό θα σήμαινε ότι δεν το θέλουμε αυτό. Όχι, θέλουμε να προχωρήσουμε σε όλα τα μέτωπα και μόνο μπορούμε να έχουμε βελτίωση αν έχουμε περισσότερα. Και τα κράτη-μέλη θα θέλουν να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όχι γιατί τα κράτη-μέλη θα πει δεν μπορείτε να λάβετε αυτά τα χρήματα, αλλά γιατί θα είναι καλύτερο ε, σε ό,τι αφορά την απόκτηση πόρων. Τώρα να συζητήσουμε τα ποσά, να το συζητήσουμε και να κάνουμε πιο ξεκαθαρή τη διαφορά. Όμω νομίζω ότι αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά στο συζητήσουμε περισσότερο συνάντηση των σκιωδών. Σε ό,τι αφορά τώρα κάποια άλλα θέματα, η επαναγκατάσταση, κύριε Λένερ, δεν θα είναι η μόνη λύση για ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Είναι ένα στοιχείο, αλλά είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο που μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να συμμετέχουμε στι παγκόσμιε ανάγκε επαναγκατάσταση τη υπερσαρμοστία μπορούμε να είμαστε λοιπόν ένα παγκόσμιο παίκτη. Τώρα, ναι, κάποιε χώρε είναι διστακτικέ. Όμω ήταν λίγε χώρε ε, που έλαβαν του περισσότερου πρόσφυγε το 2015, Γερμανία, Σουηδία και κάποιε άλλε. Για τη Σουηδία, παραδείγματο χάρη, ο στόχο που έχω θέσει δεν σημαίνει κάποια αλλαγή, σημαίνει 5.000. Αυτό είναι. Μπορεί να το θέσει κανεί και έτσι για την οικογενειακή επανένωση. Δεν είναι λογικό να έχουμε οικογενειακή επανένωση σχετική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε ταυτόχρονα ένα παράλληλο σύστημα όπου θα γίνεται και εκεί η οικογενειακή επανένωση. Γι' αυτό τα έχω ξεκαθαρίσει αυτά. Θα επανέλθω στα θέματα που έθιξε η Κομισιόν. Δεν είμαι κατά του να δούμε την επανεγκατάσταση στρατηγικά, όμως τι σημαίνει, σημαίνει ότι υποστηρίζεται καταστάσεις όπου έχεις κάποιους πρόσφυγες που χρήζουν προστασίες, έχετε μια χώρα φιλοξενίας που κάνει μεγάλη προσπάθεια να διατηρήσει την σταθερότητα και την ασφάλεια για τους ανθρώπους και αν ε, βγάλετε κάποιους ανθρώπους μπορείτε να σταθεροποιήσετε την κατάσταση. Αυτό είναι ε, από στρατηγική σκοπιά. Δεν είναι ότι θα χτίσουμε φράκτες ε, εδώ ή θα κάνουμε άλλα πράγματα η ανθρωπιστική πτυχή πρέπει να διασφαλιστεί. Τώρα το θέμα στην καταχώρηση στο ΣΥΣ και τα λοιπά. Ξέρω ότι μας πιέζει ο χρόνος, αλλά θέλω να πω το εξή. Έχουμε πάρα πολλές διαπραγματεύσεις ταυτόχρονα και οι συνάδελφοι στη Eurodac το ξέρουν. Και φυσικά έχουμε και τους μερίς διαλόγους ε, για τον οργανισμό ασύλου. Προτείνω ότι η καταχώρηση στο Eurodac ε, να μην γίνεται πριν να έχουν οι άνθρωποι μια θετική απόφαση. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ασφάλεια, αλλά όλες οι χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ουσιαστικά έχουν ασφάλεια σήμερα και τα έγγραφα που έχουν οι άνθρωποι. Σας είπα πώς λειτουργεί. Είπα ότι η αρμοστία δίνει ε, έγγραφα στα κράτη-μέλη, έχουμε και τη δική τους αξιολόγηση ότι πρόκειται για ένα πρόσφυγα που χρειάζεται διεθνή προστασία. Έτσι λοιπόν, σε ό,τι αφορά την τεκμηρίωση, ήδη λειτουργεί το σύστημα. Όμω, τι κάνουμε όταν οι άνθρωποι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε εκεί. Και είχε και ο κύριος Λουιμίσελ προτάσει σχετικά. Θα ολοκληρώσω εδώ. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Κιώδης και με άλλους συναδέλφους στην Επιτροπή Είμαι διαθέσιμη και εγώ και το γραφείο μου και πριν από τις 25 Απριλίου που έχουμε τη συνάντηση των σκιωδών. Παρακαλώ όμως μη διστάστε να έρθετε σε επαφή μαζί μου για να συζητήσουμε συγκεκριμένα <coughs> σημεία της έκθεσης ή το σύνολό της αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Malin. And... Ευχαριστώ πολύ, Μάλιν, ε, αλλά και τα μέλη. Πιστεύω ότι ήταν ένας ε, άκρος επικοδομητικός ε, διάλογος για να καταλάβουμε, μεταξύ άλλων, ότι η μετεκατάσταση διαφέρει με άλλα ε, ζητήματα και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε μια ε, πολύ καλή πολιτική ναι, για αυτό και το ότι ε, δεν γίνεται να έχουμε ένα περιορισμένο πλαίσιο. Ήταν μια πολύ καλή συζήτηση, ακόμα και τα σημεία τα οποία ανέφερε η κυρία Ντεπρή ήταν πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ τόσο ε, την εισηγήτρια όσο και τους ε, σκιώδε και τους συναδέλφου που έλαβαν τον λόγο. σα. ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να περάσουμε τώρα ε, στο ζήτημα του Δουβλίνου και αντί να χάσουμε χρόνο με την εισαγωγή μου θα έλεγα να περάσουμε κατευθείαν στην γνωμοδότρια, στην εισηγήτρια, κυρία Βίλξτρομ σε ευχαριστώ πολύ Κλωτ. Ε, ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους. Ε, επειδή την τελευταία φορά που παρουσίασα την γνωμοδότησή μου μίλησα πολύ, αυτή τη φορά θα συζητήσουμε τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει και στη συνέχεια θα συζητήσουμε τις διάφορες ε, προτάσεις. Αρχικά θα ήθελα να σας πω ότι ε, οι τροπολογίες εκφράζουν όλο το ε, πολιτικό εύρος της, του Ευρωκοινοβουλίου. Αρχικά όμως υπάρχει μια ξεκάθαρη πορεία πάνω σε αυτό. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πλειοψηφία που υποστηρίζει ένα αυτόματο σύστημα διορθωτικής μετεκατάστασης και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε ενωμένοι πάνω σε αυτό. Επίσης πιστεύω ότι ένας μεγάλος αριθμό ε, των τροπολογιών ε, θα, ε, θα υποστηρίξουν την αρχική μου έκθεση, όμως θα πρέπει να βρούμε συμβιβαστικές, οι οποίες θα έχουν την υποστήριξη μιας μεγάλης πλειοψηφίας τόσο στην Επιτροπή όσο και στην Ολομέλεια, το οποίο για πολιτικούς λόγους είναι πολύ σημαντικό. Υποχρέωση και ε, τιμή μου θα ήταν να ε, έχουμε αυτές τις ε, συμβαβιστικές ε, και τις καταλήξουμε σε αυτές από κοινού για να είμαστε ενωμένοι. Θα ήθελα επίσης ε, να επαναλάβω ε, τους ε, σκοπούς μου. Αρχικά είναι να υπάρξει μια ισορροπία και να υπάρξει μια, ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει κατά τόπους. Το έχω εξετάσει με ΜΚΟ, με τα κράτη-μέλη, με ειδικού το οποίο θα μπορέσει να διατηρήσει αυτήν την συνεκτική προσέγγιση την οποία σας παρουσίασα δεδομένη ε, τη πολυπλοκότητα του φακέλου νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι οι συμβαστικέ πάνω στι οποίε θα καταλήξουμε θα ε, διασφαλίσουν ότι το σύστημα θα διατηρήσει αυτή την ισορροπία και την συνοχή και θα λάβει ε, υπόψη και προτάσει από άλλου συναδέλφου. Θα πρέπει να είναι ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί και θα αλλάξει την πραγματικότητα κατά τόπου και φυσικά αυτό ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να είναι μια ευρωπαϊκή ανταπόκριση στα όσα ε, ουσιαστικά είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση, διότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει από μόνο του. Επίσης, το σύστημα θα πρέπει να κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη των ε, Ευρωπαίων πολιτών, των κρατών μελών, αλλά και των προσφύγων, των ετούντων ασύλου, οι οποίοι θα πρέπει να νιώθουν ότι τους λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας ε, και τους αντιμετωπίζουμε ισότιμα όπου και αν ε, βρίσκονται και όπου και αν αξιολογούνται τους. Αυτό λοιπόν θα απαιτήσει ε, προσέγγιση στην πληροφοριοδότηση ε, αλλά ταυτόχρονα ε, και ξεκάθαρους κανόνες σχετικά με το ποιο κράτος μέλος ε, θα φέρει την ευθύνη ε, για την ε, επεξεργασία της αίτηση ασύλου και το σύστημα δεν θα πρέπει να δημιουργεί δυνατότητες ή κίνητρα για τους ετούντες να παρακάμψουν το σύστημα ή να χαθούν από το ραντάρα. Και ο ένας λόγος είναι για την προσωπική τους ασφάλεια. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να εξαφανιστείς μέσα στην Ευρώπη και ιδιαίτερος όταν μιλάμε για ασυνόδευτους ενήλικες ε, γνωρίζουμε ότι δεκάδες χιλιάδες παιδιά εξαφανίζονται στην Ευρώπη. Μπορώ λοιπόν να σας πω ότι δεν θα είναι εύκολο. Έχουμε λάβει ε, περί τις χίλιες τροπολογίες, όμως κανένας δεν μας υποσχέθηκε ότι η πολιτική ζωή ε, είναι εύκολη. Θα είναι δύσκολο λοιπόν όμως ε, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να δείξει τόσο στους πολίτες όσο στις κυβερνήσεις της Ευρώπης ότι όταν συνεργαζόμαστε και μένουμε ενωμένοι τότε μπορούμε να βρούμε και είμαστε ικανοί να βρούμε κοινέ ε, λύσεις ε, που λειτουργούν και αλλάζουν την πραγματικότητα κατά τόπους. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να συνεργαστούμε, να είμαστε προσεκτικοί με τις λεπτομέρειες ε, για να μπορέσουμε να ε, διατηρήσουμε τη συνοχή του κειμένου. Είμαι πεπισμένη ότι θα βρούμε ε, δρόμο να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, θα το κάνουμε από κοινού. Αυτή τη στιγμή ακολουθούμε διαφορετικές πορείες, όμως όμως γνωρίζουμε ότι ε, δεν έχουμε τεράστια εμπόδια ε, να ε, υπερκεράσουμε, οπότε τα μεγαλύτερα εμπόδια που θα έχουμε θα είναι η αντίσταση από το Συμβούλιο και γι' αυτό το λόγο από πολιτικής άποψης είναι σημαντικό να βρούμε τον τρόπο να προχωρήσουμε προς τα εμπρός και να παραμείνουμε ενωμένοι. Αυτό είναι το κλειδί, διότι τότε το κείμενό μας ε, και η προσέγγιση μας αυτή θα ε, δώσει ε, όθηση στο Συμβούλιο ώστε να κινηθούν και αυτοί όπως κινούμαστε εμείς. Κλείνοντας λοιπόν θα ήθελα να δώσω μια θετική χρειά. Τα πάντα είναι δυνατά και η πολιτική είναι η τέχνη του δυνατού. Σας ευχαριστώ πολύ. μπορείτε να ε, χειροκροτήσετε. Ε, θα ελπίζα και άλλοι να το έκαναν, όμως ο λόγος για τον οποίο ε, δεν το κάνουν όλοι είναι επειδή αντιλαμβανόμαστε το πόσο δύσκολο είναι το έργο που πρέπει να γίνει. Ξέρω, τουλάχιστον από τη δική μας ομάδα, πόσο σκληρή δουλειά γίνεται. Ας περάσουμε τώρα στους σκιώδεις και περνάμε με την κυρία Μουσουλίνη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Εμείς είπαμε ήδη ότι θεωρούμε το κείμενο έτσι όπως ε, τροποποιήθηκε από την εισηγήτρια μία βέλτιστη βάση για τις διαπραγματεύσεις. Σίγουρα υπάρχουν κάποια σημεία που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν. Όπως και τις προάλλες, εγώ αναφέρθηκα στην ελληνική και στην ευελιξία που περιλαμβάνεται στο κείμενο, είτε ε, από την πλευρά του ετούντος ε, που ζητά μεγαλύτερη ευελιξία, το αρμόδιο κράτος μέλος. Εγώ θα ήθελα σήμερα να σταθώ στα σημεία που αφορούν την ασφάλεια, γιατί αναφέρθηκαν και αυτά από πολλούς συναδέλφους. Εγώ δεν ε, ε, θα είμαι εδώ, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στις Standard Operating Procedures, ε, στις ε, πρότυπες ουσιαστικά ε, διαδικασίες ε, που χρησιμοποιούνται μεταξύ χωρών όπως η Ιταλία και η Ελλάδα. Ενώ στο εσωτερικό, παραδείγματος χάρη στα hot spot που έχουμε στην Ιταλία, αλλά όχι σε άλλα κράτη-μέλη, εμείς έχουμε μία πρώτη σειρά διαδικασιών ασφαλείας όπως είναι η συνέντευξη, η λήψη φωτογραφίας, ένα βιοχολάκι με το νούμερο και τα δακτυλικά αποτυπώματα θα σταματήσω εδώ και θα κάνω στη συνέχεια μια παρένθεση, που είναι η πρώτη φάση, πριν από το Δουβλίνο λοιπόν. Εμείς αυτό κάνουμε ως κράτος μέλος, όμως δεν το κάνουν άλλα κράτη-μέλη γιατί δεν έχουν αυτό το σύστημα. Το σύστημα αυτό όμως στην Ιταλία δεν ε, ρυθμίζεται από νόμο. Όπως ε, ξέρετε, εμείς ε, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε εδώ το Δουβλίνο, γιατί ε, δεν υπάρχει πραγματική υποχρέωση να λαμβάνονται τα δακτυλικά αποτυπώματα δύναμη του Δουβλίνου. Αυτό σε ό,τι αφορά τώρα τις πληροφορίες. Εμείς ε, δεν έχουμε λοιπόν την υποχρέωση να λαμβάνουμε τα δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά όσοι θέλουν να ενταχθούν ε, στο Δουβλίνο και να καταθέσουν αίτηση ασύλου, ουσιαστικά έχουν την υποχρέωση να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν ας είμαστε προσεκτικά σε αυτό, γιατί κατόπιν η διαδικασία, ε, ε, έγινε διαδικασία επί κατά της εταιρείας επειδή δεν λαμβάνεται τελικά αποτυπώματα, όμως δεν είναι υποχρεωτικό, δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να το λέει αυτό. Τώρα, έναντι όλων αυτών, εγώ έχω προτείνει μία σειρά τροπολογιών δεν ε, έχω καν τροποποίηση και όπου συμφωνώ με την εισηγήτρια για να μην επαναλαμβάνουμε εκ νέου έννοιες επί των οποίων συμφωνούμε, αλλά παραδείγματο χάρη για την επιταχυμένη διαδικασία εμείς θέλουμε να τη διατηρήσουμε και όταν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας. Δηλαδή, υποχρεωτικό χαρακτήρα για τι χώρε όπου κατατίθεται η αίτηση, δηλαδή το κράτο μέλο στο οποίο ε, γίνεται η αίτηση να εφαρμόσει την επιταχυμένη διαδικασία πριν να εφαρμοστούν τα κριτήρια του Δουβλίνου σε όσους θεωρεί ότι μπορεί να θέτουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη του κράτους μέλους. Όταν ένα κράτος υποδοχής εφαρμόζει τη διαδικασία ασφαλείας γίνεται αυτόματα αρμόδιο κράτο μέλο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουμε αυτή τη διάκριση μεταξύ του κρατου μέλους υποβολής της αιτηση και αρμόδιου κρατου μέλους. Θέλαμε στη συνέχεια να καταστήσουμε πιο υπεύθυνη τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Άσυλο και τις ε, μεταφορές, ακόμη και τις ακούσιες μεταφορές. Γιατί ξέρετε ότι μετά από τέσσερις εβδομάδες ο ετών περνά από το αρμόδιο κράτος μέλος ε, σε κράτος μέλος που έχει αναλάβει την ευθύνη σε ακούσια βάση και χωρίς να έχει λες επασέ. Μπορεί να παρουσιαστεί μετά από τέσσερις εβδομάδες ε, στο αρμόδιο κράτος μέλος, αλλά μπορεί και να μην παρουσιαστεί. Αυτό είναι μια επιλογή που υπάρχει. Έτσι λοιπόν η μεγαλύτερη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασύλου και Μεταφορών θα μας δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια καθώς και η δυνατότητα οι αρχές των κρατών μελών να μπορούν να διαβουλευτούν τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον ενιαίο αριθμό, με τον αδικό αριθμό καταχώρησης έτσι ασύλου. Πάντοτε για λόγους ασφαλείας, εμείς θέλαμε να αφήσουμε και αυτή την τροπολογία. Κατά τα λοιπά, εμείς έχουμε υποβάλει άλλες τροπολογίες για τη μεταβατική περίοδο, για τα υπόλοιπα λοιπόν ε, κράτη-μέλη που θέλουν ε, τη μείωση από τα 5 στα 3 χρόνια και τη μεταφορά των ομάδων από το 30 να πάμε στο 15 για να έχουμε καλύτερο έλεγχο. Κατόπιν έχουμε και τον ορισμό της οικογένειας εδώ. Καθώς εμείς εξετάζουμε αν εντάσσονται ε, στο Δουβλίνο, εντάσσονται στο Δουβλίνο ή σε άλλη νομοθεσία η έννοια της οικογένειας, σίγουρα αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση γιατί η Κομισιόν ε, εισάγει εντός του Δουβλίνου τους αδελφούς και τις αδελφές. Ε, θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια ευρεία συζήτηση γι' αυτό. Εμείς είμαστε ανοιχτοί όμως θα πρέπει να συζητήσουμε την έννοια του οικογενειακού πυρήνα. Όμως αυτό θα πρέπει να καθοριστεί. Γιατί αν ξεκινήσουμε με το Δουβλίνο, κατόπιν θα περάσει και σε όλες τις άλλες νομοθεσίες. Και θέλω να αναφερθώ και στο θέμα των ανηλίκων. Υπάρχει μια συζήτηση. Εγώ θα θέσω μια τροπολογία για το γεγονός ότι πάντοτε ως κύρια αρχή θα πρέπει να φροντίζουμε για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και θα πρέπει γι' αυτό να μεταφέρουμε όσο δυνατόν λιγότερο τα παιδιά από κράτο μέλο σε κράτο μέλο. Γιατί εξαφανίζονται, γιατί δεν έχουμε ακόμη τα δακτυλικά αποτυπώματα για ανθρώπου κάτω των 18 ετών, εκτό αν αλλάξει Eurodac και μπορούμε να βάλουμε ήδη ότι από τα 6 έτη στου ανηλίκους μπορούμε να παίρνουμε τα αποτυπώματα. Όμω τώρα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εμπνευσιμότητα για του ανηλίκους. Γιατί? γιατί αν ο ανήλικο ε, ε, κάποιο διαφορετικό κράτος ε, μέλος μεταφερθεί, τότε αμέσως θα πρέπει να του οριστεί επίτροπος. Α, πάντοτε, όπως σας είπα, προς το βέλτιστο συμφέρον ε, του παιδιού. Αν αποφασιστεί στη συνέχεια να μεταφερθεί σε άλλο κράτος μέλος, είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχει επιβράδυση της διαδικασίας υποδοχής, ένταξης, ε, της ε, εφαρμογής των δικαιωμάτων που πρέπει να απολαμβάνει ο ανήλικος. Καθώς υπάρχει μεταφορά από κράτος μέλος σε άλλο, μπορεί να συμβεί και να εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Έτσι λοιπόν, εγώ συμφωνώ ότι είναι καλό σημείο αφετηρίας γιατί υπάρχει αυτή η ομάδα multitasking, όμως το αυτόματο δίκτυο κάπως με ανησυχεί και γιατί θα υπάρξει επιβράδυση των ε, αυτόματων διαδικασιών ένταξη για τον ανήλικο και επειδή έχουμε μικρή ανιχνευσιμότητα. Έτσι λοιπόν, ε, να έχουμε λιγότερες μετακινήσεις για τους ανηλίκους, νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια εγγύηση για το ότι θα έχουμε καλύτερη κυδαιμονία, καλύτερη επιτροπία για αυτήν την ε, πολύ ευάλωτη κατηγορία, την πιο ευάλωτη. Εντάξει, λεσάντρα, ναι, ναι, τα είπα, φτάνει. Πρέπει να τελειώσω. Ναι, πρέπει να τελειώσω. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε και μισή την όλη συζήτηση και με τόσες τροπολογίες καταλαβαίνω ε, ότι είναι σημαντικό ότι θέλετε να αναφέρετε τα πάντα όμως θα πρέπει όλοι οι σκιώδεις να μιλήσουν πριν τις 11.30 και συγγνώμη που σας διακόπτω. Για τους σοσιαλιστές, ε, Έλλη, είστε σκιώδεις. Κοιτάξτε, πρόκειται για την έκθεση για το Δουβλίνο. Το ξέρω ότι όλοι μπορούν να μακρηγορήσουν, αλλά σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδελφούς ε, για τη συνεισφορά τους ε, και θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Βίκστρομ για τη δουλειά της και τις προσπαθίες της. Θέλω να παρουσιάσω τη δική μας θέση. Όλη η προσέγγιση των τροπολογιών μου βασίζεται στην εξή βασική αρχή. Άνθρωποι που φεύγουν να γλιτώσουν τον πόλεμο και τη δίωξη δεν κατευθύνονται προς ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, αλλά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ευθύνη, να δράσει αλληλεγγύα και επίσης να αναλάβει τις ευθύνες της για το άσυλο, έτσι όπως προβλέπεται στα άρθρα 78 και 80 των συνθήκων. Το ήδη επανειλημμένος και με μεγάλη πλειοψηφία έχει ζητήσει για μια κοινή ευρωπαϊκή λύση την οποία χρειαζόμαστε. Για να είμαστε συνεπείς με ό,τι ψηφίσαμε λοιπόν στο ψήφισμα το Απριλίο του 2016 που ζητήσαμε να ξεπεράσουμε τα κριτήρια της πρώτης ε, χώρας εισόδου προς την αλήψη ευθύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαγράψαμε την αρχή της πρώτης χώρας ε, εισόδου ως ε, αρχή του συστήματος του Δουβλίνου. Τώρα για το κατόφλι, επειδή ε, ουσιαστικά δέχεται μέσω στη λογική της πρώτης χώρας εισόδου και αναπτύξαμε ένα σύστημα που βασίζεται σε μια ιεραρχία κριτηρίων και σε, μια, ένα κεντρικό και μόνιμο ε, μηχανισμό κατανομής, ο οποίος ε, λαμβάνει υπόψη ε, τους, τις συνδέσεις που μπορεί να έχει ο ετών με κάποιες χώρες. Επίσης, η έλεγχη μη παραδεκτού ήταν πολύ επικίνδυνη και καταργήθηκαν, συμφωνώ και με την προτεραιότητα που δίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία στην οικογενειακή επανένωση, κυρίω ό,τι αφορά του ανήλικου. Προτείνουμε και διεύρυνση τη έννοια τη οικογένεια, πέρα από αυτό που προτείνει την Κομισιόν, για να αντικατοπτρίσουμε καλύτερα την πολύπλοκη πραγματικότητα των οικογενειακών δεσμών των ετούντων. Δεν υποστηρίζουμε την προσέγγιση κυρώσεων που υποστηρίζει η Κομισιόν και προτείνουμε ε, να δίνουμε κίνητρα ε, για την συμμόρφωση και να μην δώσουμε κίνητρα για τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Επίσης, ε, σε σχέση με τους περιορισμούς στην προσφυγή και την ρήτρα διακριτικής ευχαίρειας, δεν τα υποστηρίζουμε. Έχουμε διαγράψει τη συνεισφορά οικονομικής αλληλεγγύης γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αγοράζει κανείς την ελληνική από τα κράτη-μέλη και να νοηματοκοποιεί τα ανθρώπινα δικαιώματα θέλουμε περισσότερες δικλείδες ε, για τους ε, ε, ανηλίκους και προστατεύουμε τα δικονομικά δικαιώματα των ετούντων. Τώρα πώς θα λειτουργήσει το σύστημα και το δίνουμε αυτό συνεισφορά στη δουλειά που έχουμε να κάνουμε στις ε, συναντήσεις των σκηνών. Καταρχήν, ε, καταχώρηση στην πρώτη χώρα, την ελαφρά διαδικασία οικογενικής επανένωσης, τα άλλα κριτήρια του Δουβλίνου, όπως και η δυνατότητα χορηγίας, sponsorship, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Καναδά. ουσιαστικά να προ μία οργάνωση που θα πλήρει κάποιες προϋποθέσεις να αναλάβει τη φροντίδα κάποιου ετούντα και αν τα κριτήρια αυτά δεν ισχύουν, η ευθύνη θα καθορίζεται από έναν κεντρικό μηχανισμό κατανομής που καταρχήν θα εξέταζε τους ε, δεσμούς ε, ε, που μπορεί να έχουμε τη χώρα, το σχάρι, τις γλώσσες που μιλάει, αν έχει κάποιο ακαδημαϊκό τίτλο ή αν έχει συγγενείς. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτοί οι δεσμοί, γιατί είναι πιο εύκολο να ξεκινήσουμε τους ανθρώπους που έχουν μια σύνδεση με τη χώρα και δεν είναι πιο εύκολο να ενταχθούν στην κοινωνία των πολιτών παρά να περιμένουμε την αυτόματη κατανομή. Επίσης, ένα περαιτέρω κίνητρο θα μπορούσε να είναι ότι αφαιρούνται, αφαιρείται το κόστος ε, αν υπάρχουν αυτοί οι σπόνσορες. Ε, αν όμως δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, θα πρέπει να ισχύει ο αυτόματος μηχανισμός και να επιτρέπεται ε, ουσιαστικά να ε, μπορούμε να αναφερόμαστε στα έξι κράτη-μέλη που είναι μακριά από το να πετύχουν το στόχο τους δύο περιπτώσεις δεν ε, θα μπορεί να γίνει. Τότε παραδείγματο ε, χάρη αν δώσει ψεύτικο όνομα οικογενειακού δεσμού ο ετών ή αν δεν έχει εγγραφεί στην ε, πρώτη χώρα εισόδου και έχει προβεί σε δευτερογενή μετακίνηση. Στις δύο αυτές περιπτώσεις ο μηχανισμός κατανομής θα γίνεται αυτόματα και θα κατανέμεται ο ετών σε κάποιο κράτος αυτόματα. Θέλουμε λοιπόν να εξαλείψουμε τα κίνητρα για δευτερογενείς μετακινήσεις ε, και να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και δίκαιο σύστημα του Δουβλίνου. Εμείς προσπαθήσαμε με τις τροπολογίες μας να δείξουμε ότι ένα άλλο Δουβλίνο είναι εφικτό. Ένα σύστημα το οποίο ε, δεν τιμωρεί τα κράτη-μέλη, ούτε τα βαρένα βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνω έκκληση λοιπόν σε εσάς συνάδελφοι. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο κανονισμός του Δουβλίνου είναι υπό αναθεώρηση. Μπορούμε μπορούμε τελικά να το φτιάξουμε μπορούμε να δράσουμε υπεύθυνα όταν το Συμβούλιο δεν το κάνει και νομίζω ότι θα πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι και να διορθώσουμε την τροπιαστική θέση Συμβουλίου για να με ισχυρή βουλή να δείξουμε ότι ναι, από κοινού μπορούμε να τα καταφέρουμε και τελικά αν όλοι τη μοιράζονται αυτή την προσπάθεια θα είναι βιώσιμη για όλους. Σε αυτές τις δύσκολες μέρες δεν θέλουμε μόνο ένα αποκλεισματικό σύστημα του Δουβλίνου, αλλά πέρα από αυτό πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας γιατί χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν προκλήσει που αντιμετωπίζουμε είναι προκλήσει και παγκόσμιε και κανένα κρατός μέλο δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο του. Πρέπει να σώσουμε την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και ανυπομονώ να συνεργαστώ με όλου σα στη συναντήση των σκιωδών. Ευχαριστώ πολύ και για το ECR ε, έχουμε τον κύριο Ντάλτεν. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σεσίλια και τους Κιώδης για το ε, έργο που έχουν κάνει. Θα ήθελα αρχικά όμως ε, να εξηγήσω μερικές από τις δικές μας ε, τροπολογίες. Ε, αφενός θέλουμε να υπάρξει ευελιξία στο κείμενο, ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να δεχθούν ετούντες οι οποίοι θέλουν να μεταβούν σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, όμως αυτό θα πρέπει να αποφασίζεται από τα κράτη-μέλη Επίσης θα είναι καλύτερο εάν ε, τα ε, κράτη-μέλη εθελοντικά ε, δηλώσουν ότι θέλουν να λάβουν πρόσφυγες αντί να εξαναγκαστούν, διότι με αυτόν τον τρόπο οι πρόσφυγες θα νιώθουν πιο, πιο ευπρόσδεκτοι και δεν θα έχουν την ανάγκη να πάνε σε άλλη χώρα. ή ε, ε, σε περίπτωση που έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν κράτο, κράτος μέλους, τότε υπάρχει ο κίνδυνος ε, να κάνουν το ταξίδι, όσοι κάνουν το επικίνδυνο ταξίδι, να έχουν την λαθασμένη εντύπωση ότι θα μπορούν να επιλέξουν το που θα πάνε με αποτέλεσμα να παίρνουν σοβαρούς κινδύνους για να φτάσουν τις εκθέσει της Ευρώπης και αυτό δεν είναι ένας λογικός τρόπος να προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης θα υποβάλω τροπολογίες για να δώσω έμφαση στην ποιότητα ταχύτητα ε, των ε, ε, διαδικασιών, ούτω ώστε να παραμένουν ενημερωμένοι καθ' όλη τη διαδικασία αλλά και τι υποχρεώσει τους και νομίζω ότι είναι, υποχρεωτικό, είναι αναγκαίο να ε, έχουμε ε, δυνατότητες, ε, να εξετάζεται η δυνατότητα έγκρισης από την πρώτη χώρα όπου εισάρχονται για να μην υπάρχει πίεση στο σύστημα και να μην περιμένουν οι ετούντες για πάρα πολύ καιρό μέχρι να εκδοθεί η απόφαση. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το συμφέρον των παιδιών και αυτό σημαίνει, ότι θα πρέπει να έχουμε ευελιξία όσον αφορά την επιστροφή των ασυνόδευτών στην πρώτη χώρα εισόδου σε περίπτωση που αυτό είναι προς το συμφέρον συμφέρον δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου θα δίνουμε το κίνητρο στους ανήλικες ε, να ε, ταξιδεύουν μόνοι τους σε όλη την Ευρώπη ε, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από τους διακινητές. Επίσης όσον αφορά τον μηχανισμό ανακατανομής δεν έχουμε αλλάξει άποψη, στηρίζουμε το ίδιο και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι εθελοντικός και να εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη ως κατευθυντή και, και όχι ω υποχρέωση και δεν θα πρέπει ε, τα κράτη-μέλη να ε, υποχρεούνται να αποδεχθούν έναν αόριστο αριθμό ετούντων. Ε, αν υποχρεώσουμε κάτι τέτοιο και να, ασκούμε, ε, να επιβάλλουμε ποινέ, δεν είναι ο σωστό τρόπο προώθηση τη ελληνική, αλλά και ούτε ο σωστό τρόπο για να νιώθουν ευπρόσδεκτοι πρόσφυγε όταν φτάνουν εδώ πέρα. Έχουμε ευρεία συμφωνία όσον αφορά τι ποινέ, διότι κάτι τέτοιο δεν θα εθαρρύνει την ελληνική μεταξύ των κρατών μελών και επίση θα ήθελα να τονίσω ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε απλά οικονομικές ε, κυρώσεις, ε, διότι ε, κάτι τέτοιο δεν το υποστηρίζουμε εμείς. Όπως και να έχει όμως, ευχαριστούμε τη Σίλια για το έργο που έχει κάνει ως τώρα και προσβλέπουμε στη συνεργασία που θα έχουμε, ούτως ώστε να έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε. Ο επόμενο ομιλητή είναι ο κύριος Ζαν Λαμπέρ. Ευχαριστώ πολύ. όσον αφορά τη δική μας ε, προσέγγιση ε, δεν θα ε, υποβάλουμε τροπολογίες στα πάντα, όμως ορισμένα θέλουμε να τα τονίσουμε και το ένα εξ αυτών είναι το θέμα των ποινών σε περίπτωση που δεν τηρούν τους κανόνες υποδοχής, διότι εδώ εξετάζουμε κάτι όπου προσπαθούμε να συνεργαστούμε και με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα Επίσης πιστεύω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ενώ έχουμε ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία ε, έχουν ορισμένη πίεση, αυτό έχει αλλάξει και ίσως να αλλάξει και στο μέλλον. Έτσι λοιπόν τα κράτη-μέλη όταν εξετάζουν το συγκεκριμένο και όταν το κάνουμε και εμείς αυτό, θα πρέπει να λαμβάνουμε όλο αυτό υπόψη μας ε, και να μην ε, αναλογιαζόμαστε μονάχα την παρούσα κατάσταση. Διότι κάποια κράτη-μέλη τα οποία αντιστέκονται σε μέτρα αλληλεγγύη ίσω ίσως να έχουν ανάγκη αυτών ε, στο μέλλον και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το τι ίσως να συμβεί μελλοντικά. Όσον αφορά τις ε, τροπολογίες που έχουμε καταθέσει θα αναφέρω ε, δύο-τρεις εξ αυτών. Ε, μία αφορά το ζήτημα τον ορισμό της οικογένειας. Ακούω το τι λένε ορισμένοι ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε και να έχουμε μια κοινή προσέγγιση πάνω σε αυτό. Από την άλλη όμως έχουμε τις συνθήκες υποδοχής και η συγκεκριμένη οδηγία είναι μια οπότε δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τον ορισμό της οικογένειας. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν να μην, να μπούμε σε μια σειρά αποφάσεων εξαιτίας μιας ε, πρότασης αναδιατύπωσης ε, την οποία δεν μπορούσαμε ε, να επεξεργαστούμε στο, στον πυρήνα της. Τώρα όσον αφορά τους ετούντες ασύλου, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει, έχουν αντιμετωπίσει συγκεκριμένες καταστάσεις και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό ε, και ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε πέραν αυτού όσον αφορά τον ορισμό της οικογένειας. Ένα ε, θέμα το οποίο έχουμε θέσει αφορά το ερώτημα της της, ε, του γάμου ε, εάν μπορεί κάποιος ε, να επανενωθεί με την σύζυγο ή τον σύζυγο εάν είναι σε ένα κράτος μέλος που δεν έχει αναγνωριστεί. Τι γίνεται εκεί πέρα θα πρέπει να εξετάσουμε τους οικογενειακούς δεσμούς και να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Επίσης, θα πρέπει να ε, διευρύνουμε ε, τους δεσμούς πέραν της οικογένειας, διότι πιστεύουμε ότι οι ετούντες ασύλου δεν ε, λαμβάνουν απλά ε, βοήθεια, αλλά έχουν και έναν συγκεκριμένο σκοπό. Αν είμαστε σοβαροί λοιπόν ε, για την ενσωμάτωσή τους ε, και να διάγουν ένα βίο όπου κάποια στιγμή θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις χώρες τους, τότε το ζήτημα της ενσωμάτωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι για το οποίο συζητούν έντονα τα κράτη-μέλη και κάποια από τα ζητήματα τα οποία προσφέρουν είναι που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε. Έχουμε μια σειρά τροπολογιών που αφορούν τη διευρυμένη οικογένεια, αλλά και ζητήματα όσον αφορά ε, τις, τους πολιτισμικούς δεσμούς, τη γλώσσα, ε, τους οικογενειακούς δεσμούς ε, και όλα αυτά θα πρέπει να, λαμβω, να ληφθούν υπόψη. Όλα αυτά όμως δεν... Κάποια από αυτά υπάρχουν, κάποια όχι. Και υποστηρίζουμε την ιδέα του να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης σε ομάδες παρά να ε, διανέμονται οι άνθρωποι ε, σαν να είναι ε, χαρτιά μια τραπουλόχαρτας, μια τράπουλα. και θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην διανύμουμε τους πόρους πολύ αραιά σε ανθρώπους διαφόρων υποβάθρων. Επίσης, το ζήτημα αφορά επίσης ε, την ε, διαδικασία ε, επανεισδοχής. Όλα τα κράτη-μέλη πρώτης εισόδου θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ έντονο έργο και με αποτέλεσμα όλος ο μηχανισμός να μην λειτουργήσει πραγματικά και γι' αυτό το λόγο δεν εξετάζουμε ένα μηχανισμό ελληνική. Επίσης έχουμε υποβάλει τροπολογίες οι οποίες βασίζονται στο ε, έργο ε, της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όπου, εξετάζουν, όπου έχουν δουλέψει με τους ετούντες ασύλου πολλά από, πολλές από τις πρώτες αποφάσεις ε, των κρατών μελών μας εφεσιβάλλονται, οπότε θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικότερα, αποτελεσματικότερα και πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και ε, τώρα η κυρία Φεράρα. Ο κύριος Κόρα που αντικαθιστά την κυρία Φεράρα. Μάλιστα αντικαθιστώ την κυρία Φεράρα. Αυτό το σημείο είναι τεχνικού χαρακτήρα και βλέπουμε τις θέσεις διάφορων ομάδων, αλλά έχει πολύ σημαντική πολιτική αξία για μια σωστή μεταρρύθμιση του κανονισμού του Διβλίνου. Πιθανόν ε, εδώ διακυβεύεται και η πολιτική αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων. Εμείς έχουμε παρουσιάσει κάποιες τροπολογίες, τις οποίες διευκρινίσαμε τις θέσεις μας ε, για τον κανονισμό αυτό. Παραδείγματος χάρη, δεν θέλουμε το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο ε, το κράτος ε, μέλος που είναι υπεύθυνο πρέπει να είναι το πρώτο κράτος μέλος ε, εισόδου και το αντικαθεστούμε με μία αναφορά στη χώρα όπου παρουσιάζεται, είναι παρόν ο ετών άσυλο. Σύμφωνα με εμά, το αρμόδιο κράτος είναι αυτό που έχει οικογένεια ο ετών και συμφωνούμε με, την διευρυμένη, ε, με το διευρυμένο ορισμό και θέλουμε μία ταχεία ε, διαδικασία οικογενικής επανένωσης, ε, παραδείγματος χάρη μέσα σε ένα μήνα να μπορεί να μεταφερθεί στο κράτος όπου ισχυρίζεται ότι έχει οικογένεια ο ετών. Επίσης, ε, αν δεν πληρούνται αυτές οι ε, προϋποθέσεις, θέλουμε να γίνεται αυτόματα η κατανομή και όχι μόνο επειδή θα έχουν καταρρεύσει τα εθνικά συστήματα και αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη. Αυτό έλειπε μέχρι τώρα και είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Ο μηχανισμός ε, μοιράζει τους ετούντες βάσει μιας κλίδας που λαμβάνει υπόψη κριτήρια όπως είναι το ΑΕΠ και ο πληθυσμός. Εμείς έχουμε προσθέσει και το ποσοστό ανεργίας για την κατανομή των ετούντων στα διάφορα κρατημέλη, πέρα από την μέθοδο που προτείνει η Κομισιόν, την αριθμητική, προτείνουμε να λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη παρουσία ε, σε κράτη του ετούντο. αν μιλά κάποιες ε, γλώσσες ε, και αν έχει πολιτιστικούς δεσμούς. Προτείνουμε τη διακοπή της καταβολής ε, των ε, κονδυλίων των ορθρωτικών ταμείων σε κράτη-μέλη που δεν συμφωνούν να συμμετέχουν στο μηχανισμό κατανομής. Γιατί διαφορετικά, αν δεν λείπει καμία κύρωση, απλώς θα φλιαρούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τη θέση της ε, εισηγήτριας Βίκστρομ, εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να δέχουμε το κύριο κριτήριο για την ε, απονομή της ευθύνης να παραμένει το, η πρώτη χώρα της ε, παράνομης ε, άφηξης, γιατί αυτό έχει οδηγήσει ουσιαστικά στην κατάρρευση ολόκληρου του συστήματος ασύλου τα τελευταία χρόνια. Το να διατηρήσουμε ένα μηχανισμό ανακατανομής που δεν είναι νόμιμο, μόνιμος, θεωρούμε ότι δεν είναι μια λύση, γιατί μειώνει το κατόφλι επί το οποίο θα πρέπει να περιοδοτείτε, όμως ε, αυτό ε, δεν ε, σημαίνει, μάλλον αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός θα πυροδοτείται όταν έχει καταρρεύσει ήδη το σύστημα τους κράτους μέλους. Κανένα κράτος μέλος ε, δεν ε, μπορεί να έχει ε, τελικά μία περίοδο μεταβατική για να φτιάξει τα συστήματά του. Τα συστήματα σύλλου υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ, πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Ήδη έχει γίνει δουλειά πάνω στην οργάνωση των συστημάτων ασύλου. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά έναν έμεσο τρόπο για να αποφύγει τις ευθύνες του το κράτος μέλος. Και αν το υιοθετήσουμε τελικά βλέπουμε τι θα γίνει όπως κάποια κράτη δεν δέχτηκαν ούτε λίγες χιλιάδες πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε την εισηγήτρια και ελπίζουμε ότι πραγματικά μετά από τόσες καθυστερήσεις και τόσες ε, αποτυχίες να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε αυτή τη φορά και να έχουμε μια συγκεκριμένη θέση που θα ακολουθήσουν και τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά θα χάσουμε οποιαδήποτε αξιοπιστία έχουμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. <coughs> Okay, thank you. Uh, now, uh, uh, we finished. Ε, ωραία, ακούσαμε ε, τους ε, σκιώδεις ε, και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Λέναρς. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ε, στενάχωρο το γεγονό ότι έχουμε τη συγκεκριμένη πρόταση, ε, διότι η αλληλεγγύη για την οποία έχουμε ε, εκφράσει πολύ δεν υπάρχει και συμφωνώ, δεν είμαι σύμφωνο των υποχρεωτικών ποσοστώσεων επανεγκατάσταση προσφύγων ή ετών ασύλου εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω κάτι το οποίο φάνηκε τα τελευταία χρόνια είναι ότι άμα το αφήσουμε να είναι εθελοντικό δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, θα υπάρχει ισότιμη διανομή ε, ευθύνη και θα είναι αποτελεσματική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, κάτι για το οποίο έχω ερώτημα και ίσως να είναι και χαζό ερώτημα όταν αφορά την κλίδα ε, εκεί το θα πρέπει να προσθεθεί ο αριθμός των επιτυχόντων μετεγκαταστημένων ε, αναρωτιέμαι ότι αν αυτός δεν είναι και ένας ε, τρόπος ε, για να δημιουργήσουμε ένα υποχρεωτικό σύστημα επανεγκατάστασης στο εσωτερικό της Ένωσης και θα ήθελα να ακούσω και την απάντηση της Κομισιόν είναι μια υποθετική κατάσταση όπου για παράδειγμα οι πράσινοι κερδίσουν του χρόνου τις εκλογές στην Ουγγαρία και αποφασίσουν να επανεγκαταστήσουν 200.000 ε, ε, ανθρώπους στην Ουγγαρία για να ε, επιτύχουν τον στόχο τους, οι άνθρωποι αυτοί στη συνέχεια υποχρεωτικά θα αναδιανεμηθούν στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και αυτός ο μέσος όρος θα πρέπει να είναι ποσοτικός, να λαμβάνεται υπόψη όταν κάνουμε την αναδιανομή ε, και ε, θα, πρέπει, θα ήθελα να ακούσω αν θα υπάρξει μια ε, συγκεκριμενοποίηση πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ράντεφ. Η Κομισιόν είχε μια δυνατότητα τώρα για να αλλάξει την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με το άσυλο, ε, καθώς το Κοινοβούλιο το ζητά αυτό εδώ και καιρό. Θέλουμε ένα σύστημα που να ευνοεί και τους ετούντες άσυλο, αλλά και τα κρατημέλη να βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, η Κομισιόν ε, δεν παρουσίασε την κατάλληλη πρόταση. Εμείς έχουμε εισαγάγει κάποιες τροπολογίες για να ανακουφίσουμε τα κράτη που είναι στα εξωτερικά σύνορα, όπως η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιταλία, που δεν θα έπρεπε πλέον να είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία χιλιάδων ετήσιων ασύλου. Οι μετανάστες δεν ε, θα πρέπει να στέλνονται στην ε, πρώτη χώρα υποδοχής. Επιμένουμε σε αυτό. Κατανοώ την ανησυχία των υπόλοιπων κρατών ελών για τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Παρ' όλα αυτά, τέσσερις ή πέντε χώρες ε, δεν μπορούν να σηκώσουν όλο το βάρος, ενώ οι υπόλοιπε αρνούνται να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια, μάλιστα ούτε καν τεχνική βοήθεια δεν προσφέρουν. Έτσι λοιπόν θέλω να απευθύνω έκκληση στην εισηγήτρια και στους σκιώδεις εισηγητές να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα που να μπορεί να ανακουφίσει τα κράτη-μέλη που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης. Εμείς θα θέλαμε το σύστημα του Δουβλίνου να τροποποιηθεί, καθώς είναι αποτελεσματικό όταν ε, υπάρχουν πολύ μεγάλες μεταναστευτικές πιέσεις. Ευχαριστώ. Merci, Madame la επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Σμένοβα. Καταρχήν ε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βίξτρομ ε, για τη δουλειά της ε, για αυτό το δύσκολο φάκελο. Πολλές φορές στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ υπογραμμίσαμε την αναγκαιότητα μιας πλήρης επανεξέτασης του μηχανισμού του Δουβλίνου γιατί μας έδειξε η κρίση των τελευταίων χρόνων της ανεπάρκειας επίλυσης του προβλήματος. Οι διατάξεις για την ευθύνη των χωρών πρώτης εισόδου ε, ε, μας οδήγησε σε μια δυσανάλογη πίεση σε κάποιες χώρες όπως Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία. Αυτό είχε αρνητική επίπτωση στο σύστημα ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη λειτουργία της Ένγκεν. Γι' αυτό πιστεύω, μάλλον ελπίζω, ότι οι νέοι κανόνες δεν θα επαναλάβουν τα ίδια λάθη και ότι θα προβούν σε πραγματικό επιμερισμό της ευθύνης καθώς ε, προέρχομαι από μία από τις χώρες που πλήττονται, θέλω να κάνω έκκληση η γεωγραφική τοποθεσία των χωρών αυτών να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το άσυλο. Επίσης, ε, πρέπει να υπάρχει σαφήνεια για τον αριθμό των καταχωρημένων ανθρώπων. Όμως, οι χώρες της περιφέρειας δεν έχουν ε, αυτά τα νούμερα. Γι' αυτό οι χώρες της περιφέρειας θα πρέπει να ε, έχουν ένα περιθώριο αντίδρασης όταν έχουμε μαζικές αφήξεις. Το 150% που προβλέπεται για την πυροδότηση του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής είναι κάτι πολύ ψηλό γιατί προϋποθέτει την κατάρρευση του συστήματος ασύλου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ε, και μετατρέπει το μηχανισμό της ισότητας ε, ε, σε ένα μέτρο που θα καταπολεμήσει τα προβλήματα και μπορεί τελικά να είναι τόσο αναποτελεσματικό όπως και η τυχαία κατάσταση. Επίσης προτείνω στην περίπτωση που έχει απορριφθεί μια αίτηση και έχει αποσταλεί σε τρίτη χώρα ο μετανάστης η μόνιμη ευθύνη της ε, χώρας που έχει εξετάσει το αίτημα θα πρέπει να λήξει γιατί ε, διαφορετικά ε, θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για το αν ο άνθρωπος αυτός ξανακαταθέσει το αίτημά του σε άλλες χώρες. Αυτό δεν έχει λογική. Τέλος η κυρία ε, Ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως ε, το να συζητάμε, το να φτάσουμε να συζητήσουμε μια τροποποίηση των χαρισμών του Δουβλίνου ήταν ένα βήμα προς τα μπρος. Γι' αυτό δεν πρέπει να σπαταλήσουμε αυτή την ευκαιρία. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε ριζικά να αλλάξουμε τον κανονισμό του Δουβλίνου. Όμως βλέπω δυστυχώς ότι δεν ε, έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Γιατί θα ήθελα να δω μια πολύ φιλόδοξη ε, πρόταση από το Κοινοβούλιο εμείς πρέπει να δώσουμε ξεκάθαρη απάντηση και στους πολίτες αλλά και στις ε, χώρες της ε, πρώτης άφηξης. Πολλές κυβερνήσεις της Ένωσης δείχνουν έλλειψη πολιτικής βούλησης και αυτό έχει στείλει σε κρίση την ίδια τη λειτουργία του κανονισμού του Δουβλίνου και σήμερα απαιτείται ριζική αλλαγή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο και απλώς να κάνουμε μικρές τροποποιήσεις, πρέπει να αλλάξουμε ένα ολόκληρο σύστημα, να έχουμε ένα κεντρικό σύστημα. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξει μια πιο φιλόδοξη πρόταση και να εργαστεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τα κρατημέλη για να φτάσει σε αυτό το στόχο. Εγώ λυπάμαι που λέω που η αρχή της αλληλεγγύης που έχουμε ήδη στις συνθήκες μας ε, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα πλήρως και η βάση ε, να ξεπεράσουμε το Δουβλίνο ε, ποια είναι. Σήμερα βλέπουμε κρίση ελληνικής μεταξύ διάφορων κρατών μελών. Πέρσι ήδη ψηφίσαμε το ψήφισμα για την ολιστική προσέγγιση και είπαμε ότι θέλαμε ένα κεντρικό σύστημα. Εγώ παραμένω στη θέση αυτή, εμένω στη θέση αυτή να βρούμε όλες τις κατάλληλες τροπολογίες που θα πρέπει να υποστηρίξουν την πρόταση αυτή για να φτάσουμε σε ένα κεντρικό σύστημα. Σήμερα δεν χρειαζόμαστε μικρές τροποποιήσεις, περνά ο χρόνος και δεν θα μπορούμε να σταματήσουμε τη μετανάστευση. Σε τέσσερα χρόνια θα ξανάρθουμε να κάνουμε άλλη μια τροποποίηση εδώ. Θα πρέπει με κάθε τρόπο να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση καθώς ε, δεν ενισχύονται οι νόμοι μεσοδοί της μετανάστευσης, μόνο ένα αποτελεσματικό σύστημα θα μπορούσε να σώσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Πρέπει να εγγυηθούμε σε όσους χρειάζονται προστασία ότι πράγματι θα τη λάβουν, ε, όχι απλώς κατά το ίμιση. Έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη σήμερα και αυτή η ευκαιρία μας δίνεται. Δεν μπορούμε λοιπόν να την ξοδεύσουμε στο κοινοβούλιο, θα πρέπει να την αδράξουμε. Ευχαριστώ. Και ε, τώρα τελευταία αλλά όχι ε, έσχατη η κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνατε. Όλοι γνωρίζουμε τις ε, δυσκολίες αυτού του φακέλου. Και εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι αναγκαιότερο να έχουμε επικοδομητική προσέγγιση για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης και ανάληψης ευθύνης προκειμένου να υπερασπίσουμε τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μείνει κενό γράμμα, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται η έκθεση από συγκεκριμένα μέτρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, τροπολογίες που προτείναμε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αναγκαιότητα των κρατών μελών που είναι στην πρώτη γραμμή και έχουν ε, εξωτερικά σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα ήθελα να αναφέρω πέντε στοιχεία. Καταρχήν, να προσδιοριστεί το αρμόδιο κράτος για την επεξεργασία της ε, αίτηση. Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε την αρχή της ελληνικής, ε, της ε, μεταχείρισης ε, της αίτηση. Έχουμε δει ότι παρέλυσε το σύστημα όταν βασιστήκαμε στην αρχή της αρμοδιότητας του κράτους πρώτης άφηξης. Θα πρέπει να αναλυφθούν οι ευθύνες από το κράτος όπου έχει κατατεθεί έτσι, όχι από το κράτος πρώτης εισόδου. Η μόνιμη ευθύνη. Δεν είναι αποδεκτό τα κράτη-μέλη να έχουν ε, ε, την ε, ευθύνη για έναν αετούντα άσυλο, ακόμη και αν αυτός έχει εγκαταλείψει για πολύ καιρό την επικράτειά του. Έτσι λοιπόν, αν ε, εγκαταλείψει ο ετών την επικράτεια του κράτους για πάνω από τρει μήνες, θεωρούμε ότι πρέπει να μην είναι αρμόδιο το κράτος αυτό για την αιτησή του. Επίσης, για το διορθωτικό μηχανισμό. Εμείς θέλουμε να αλλάξει αυτός ο αριθμός στο 150%. Θέλω να αναφέρω τέσσερα στοιχεία επίσης. Η ρήτρα οικονομικής ελληνικής είναι μια προσέγγιση που δεν θεωρούμε ότι είναι σκόπιμη. Επίσης, εμείς ε, θέλουμε να καταργηθεί αυτή η ρήτρα της οικονομικής ευθύνης σε περίπτωση άμεσης απειλή για την ασφάλεια στα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν περιθώριο λιγμών. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τις διαπραγματεύσεις για το σύστημα εισόδου-εξόδου, όσο συνεχίζονται αυτές οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να καταλήξουμε σε, μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις σε ένα αποτελεσματικό μηχανισμό για να καταπολεμήσουμε τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Επίσης, θα πρέπει να μπορέσουμε να ελέγξουμε την ασφάλεια. Αν είναι ασφαλή ο υποψήφιο, θα πρέπει να βρούμε ποια είναι η ταυτότητά του χρησιμοποιώντα τι βάσει δεδομένων. Εγώ αυτά ήθελα να τονίσω σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Σίγουρα έχουμε πάρα, ε, πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας για να βρούμε τις κατάλληλες συμβαστικές τροπολογίες. Όμως είμαστε πεπισμένοι ότι μόνο οι κοινέ δράσεις θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την ε, σημερινή μεταναστευτική κρίση. Εμείς ε, έχουμε διανύσει μεγάλο δρόμο για να μπορέσουμε να θεσπίσουμε αυτό το σύστημα χορήγησης ασύλου. Ευχαριστούμε. Πριν δώσουμε το λόγο στην Ισχύτρια να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Παρακαλώ. Η κυρία Άννα από την Γενική Διεύθυνση Home, ο κύριος μάλλον δεν θα είναι πρόεδρος. Γενική Διεύθυνση Home. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, την κυρία Βίλστρομ, για την ε, τόσο καλή πρότασή της που παρουσίασε ήδη πριν από μερικές εβδομάδες και θέλω να ευχαριστήσω και τους και όδες εισηγητές και όλους τους ευρωβουλευτές που βέβαλαν πάνω από χίλιες τροπολογίες στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό δείχνει όχι μόνο το πόσο περίπλοκο, σημαντική είναι η ρύθμιση αυτή, αλλά και πόσο σημαντική είναι επίσης. Κάτι το οποίο είπανε πολλοί από εσά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετάει λοιπόν προσεκτικά τις τροπολογίες αυτές και προσβλέπει στην έκθεση στην οποία θα καταλήξετε εδώ στην Επιτροπή σας. Θέλω όμως να υπενθυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο περίπου, τον Απρίλιο πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση στην οποία ε, με μεγάλη ειλικρίνεια ανέφερε τις αδυναμίες του συστήματος του Δουβλίνου και του συστήματος ασύλου. Γιατί το θέμα των ροών, για το πώς έχει σχεδιαστεί το σύστημα, αλλά και πώς εφαρμόζεται το σύστημα, που δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τόσο μεγάλες μεταναστευτικές ροές, πόσο περίπλοκοι είναι οι κανόνες, ότι οι διαδικασίες κρατάνε πάρα πολύ χρόνο. το θέμα της μεταφοράς της ευθύνη που ήταν μερικές φορές δυνατό να γίνει, άλλες φορές όχι. Όλα αυτά προσθέτουν στην περιπλοκότητα και στη δυσκολία και στην αδυναμία του συστήματος, με αποτέλεσμα να στηβάζονται άνθρωποι στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε δευτερογενείς μετακινήσεις μεταξύ των χωρών μελών και σε μια κατανομή βάση του κανονισμού τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έτσι όπως έχει ο κανονισμό σήμερα δεν είναι ικανοποιητικό. Γι' αυτό και προτείναμε μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου για από πέρυσι. Εκεί προβλέπεται μια μεγάλη καινοτομία που νομίζω ότι αποτελεί και το αντικείμενο των περισσότερων τροπολογιών που προτείνει η Επιτροπή σας. Είναι και το κύριο θέμα συζήτηση στο Συμβούλιο μέχρι τώρα. Αυτή η καινοτομία είναι η εισαγωγή ενός μηχανισμού διορθωτικού που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη που έχουν τεράστιο βάρος ε, λόγω πολλών αιτήσεων ασύλου όταν φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο νούμερο που θα είναι βέβαια ανάλογο με το ΑΕΠ τον αριθμό των κατοίκων κτλ. να μπορούν τότε αυτό το βάρος να το μεταφέρουν σε κάποια άλλη χώρα. Γίνονται συζητήσεις στα υψηλότερα δυνατόν επίπεδα και ένα συμπέρασμα στο οποίο έχουμε καταλήξει, μια κοινή θέση ελπίζω να επιτευχθεί από το Συμβούλιο, θα έρθει και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση και ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το τελικό αποτέλεσμα πάντως της διαδικασίας πρέπει να είναι ισορροπημένο, ρεαλιστικό, με προβλεψιμότητα και φυσικά με δικαιοσύνη, αν θέλουμε να είναι βιώσιμο. Γι' αυτό και χρειάζονται συμβιβασμοί από όλε τις πλευρές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως πιστεύει ότι μια τέτοια ισορροπημένη λύση θα είναι αυτή στην οποία θα καταλήξουμε. Και δύο λόγια για να απαντήσω στον κύριο Λέναρτς. Ήταν η μόνη ουσιαστικά ερώτηση που ακούσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης σήμερα το πρωί. Είναι αλήθεια ότι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μερίδιο των, ε, της, κάθε χώρας ε, μέλους δεν θα αντικατοπτρίζει μόνο τον αριθμό των αιτήσεων ασύλου για τις οποίες ε, είναι υπεύθυνο το κράτος μέλο, αλλά θα υπολογίζονται και οι άνθρωποι τους οποίους σε θελοντική βάση θέλει να επανακαταστήσει. Αυτό αντικατοπτρίζει όμως το βάρος της υποδοχής ατόμων οι οποίοι χαίρουν διεθνούς προστασίας. Συγχρόνως πρέπει να υπάρχουν και κίνητρα προς τις χώρες μέλη για να προβαίνουν σε επανακαταστάσεις, όχι το αντίθετο. Οπότε θέλω να διαβεβαιώσω τον κύριο Λέναρτς ότι δεν είναι πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λειτουργήσει το σύστημα με τέτοιο τρόπο ώστε μία χώρα να επιλέγει μονομερός να επανακαθιστά έναν μεγάλο αριθμό ατόμων και μετά τα άτομα αυτά να κατανέμονται μεταξύ των υπόλοιπων χωρών μελών. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Συγχρόνως η Επιτροπή πρότεινε πρόταση κανονισμού και επαναγκατάσταση και για την τροποποίηση των διαδικασιών που να μην συμπεριλαμβάνονται σε οδηγία αλλά σε κανονισμό. Όλα αυτά μαζί όταν εγκριθούν νομοθετικά θα οδηγήσουν σε κάτι που δεν θα επιτρέπει αυτό το σενάριο το οποίο φοβάται ο κύριος Λέναρτς. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Παρακαλώ από την Μαλτέζικη Προεδρία τώρα, κυρία Μαρκής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, τους σκιώδες εισηγητέ και τους ευρωβουλευτές για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα στην υπόθεση αυτή και σας ευχαριστώ και για όλο τον προβληματισμό που προσθέτουν οι τροπολογίες. Και άλλη φορά σε συναντήσεις της Επιτροπής αυτής σας έχω εξηγήσει πώς προχωράει το έργο στο Συμβούλιο, οπότε σήμερα θα περιοριστώ για να σας πω ότι σημείωσα τις απόψεις που εκφράσατε και θα τις μεταφέρω στο Συμβούλιο για παρατέρω προβληματισμό και εκεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ωραία. Ευχαριστούμε. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε. Η Σεσίλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, συνάδελφοι, δεν με εκπλήσουν αυτά που άκουσα. Όχι. Κανείς δεν κατάφερε να με εκπλήξει από αυτά που άκουσα σήμερα. Περίεργο δεν είναι. Λοιπόν, είμαστε ενωμένοι, είμαστε μια ομάδα και θα φροντίσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες ώστε να υπάρχει συνοχή στο κείμενο και να είναι δυνατό, έντονο. Θέλω επίσης να πω στους συναδέρφους που δεν συμμετέχουν στη διαπραγματευτική μου ομάδα ότι είναι η πρώτη φορά που ο κανονισμός του Δουβλίνου αλλάζει και γίνεται ένα μέσο αλληλεγγύης. Θέλουμε όντως να διευκολύνουμε τις χώρες μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή από το βάρος που έχουν επομιστεί. Και όπως είπανε και οι σκιώδες και φαίνεται και στη δικιά μου έκθεση, πρέπει να δώσουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή απάντηση σε μια ευρωπαϊκή κρίση, σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και αυτό θα το καταφέρουμε μόνο αν μείνουμε ενωμένοι και το κάνουμε μαζί. Τώρα, για τον κύριο Λέναρτς, ο οποίος όντως κατέδειξε το πρόβλημα, λέει Μα προσπαθήσαμε με το Συμβούλιο, προσπαθήσαμε σε θελοντική βάση, όπως η Οδική για την Προσωρινή Προστασία, που ποτέ όμως δεν ενεργοποιήθηκε. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε επιτρέποντας μια δίκαια κατανομή ευθυνών μεταξύ όλων των χωρών μελών. Τροποποίησαμε για να λάβουμε υπόψη μας τις ανησυχίες των Βουλγάρων συναδέλφων, για παράδειγμα, εγώ κατέβασα το όριο για την ενεργοποίηση του μηχανισμού ή με την κατάσταση αντί και 150% που λέει πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγώ το έκανα 100%. Και θα πρέπει να μειωθεί, να γίνει 75%. Υπάρχει κάποιο περιθώριο ελιγμών. Τώρα το στοιχείο κλειδί, κατά τη γνώμη μου, και εδώ νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω εκ μέρους και των σχεδόν εισηγητών, είναι ότι θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που να είναι ουδέτερο, για να επανέλθω σε αυτό που είπε Τζιν. Σήμερα είναι η Ελλάδα και η Ιταλία, χώρε τη πρώτη γραμμή που αναλαμβάνουν το βάρο. Μπορεί να είναι η Λιθουανία ή η Πολωνία, αν κάτι συμβεί στα ανατολικά μα σύνορα, για παράδειγμα, ή στη Μέση Ανατολή, μπορεί να είναι η Κύπρο, που σε βρίσκεται ελάχιστα χιλιόμετρα μακριά από εκεί. Συνεπώ, πρέπει να προβλέψουμε, δηλαδή να μην περιοριστούμε στο πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφτηκε η πρόταση βάσει των όσων έγιναν το 2015. Μπορεί να μα περιμένουν άλλε καταστάσει. νέε, οπότε η απάντηση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που να αντέχει και να αλλάξει την πραγματικότητα επιτόπου. Διότι πρόκειται για μια δυναμία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μα, μια αποτυχία. Και έχουμε τη μοναδική ευκαιρία αυτό να το αλλάξουμε, να το αντιστρέψουμε. Η Ευρώπη το χρειάζεται. Και αυτό που διακυδεύεται είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, η ίδια αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τώρα, χάρη σε όλους εσάς θα συνεχιστεί ο διάλογος για να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για τις προσπαθίες σας, για τις τροπολογίες σας και Τώρα επιστρέψτε για τα Χριστούγεννα, λέει η κυρία Αβάστον. Πω, πω, πω τα μπέρδεψα, βιάζομαι. Πάσχα ήθελα να πω, Πάσχα. Καλό Πάσχα. Ξεκουραστείτε, εμπνευστείτε, διαβάστε καλά βιβλία και φροντίστε να επιστρέψουμε με καθαρό το μυαλό μετά τις πασχαλινές διακοπές με νέες ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ μας. Καλό Πάσχα λοιπόν σε όλους και καλές διακοπές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας. Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι το σημείο 15. Πώς θα δημιουργήσουμε έναν ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής για τους σκοπούς κοινών διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση και ανάκληση της ε, διεθνούς προστασίας. Αγαπητοί συνάδελφοι. Η συγγήτρια είναι η κυρία Σεβίγγιο. Και θα ακούσουμε και την Μαλτέζικη Προεδρία. Έχουν γίνει συναντήσεις ήδη με τους σκιώδεις συζητητές και λοιπά τους τελευταίους μήνες και έχουμε και την διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόσφατα ανακοίνωσε το Συμβούλιο την απόφασή του να σταματήσουν οι συζητήσεις για αυτό το θέμα προκειμένου να συνεχίσει η συζήτηση για ένα κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών. Είμαστε στα πλαίσια του σου διαλόγου και του κανονισμού ασύλου. Ως πρόεδρος από την ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ δεν μπορώ να εκφράσω την ε, δυσαρέσκειά μου για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν φέρει σε πέρα στις υποχρεώσεις του και τις ευθύνες του, κάτι το οποίο δεν ευθυγραμμίζεται με τις συνθήκες Υπάρχει ένα έγγραφο από το Σεβούλιο για την ε, δικιά του θέση. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην εισηγήτρια και μετά στη Μαλτέζικη Προεδρία και μετά θα δώσω το λόγο στους εισηγητέ και σε όποιον άλλον θέλει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Κυγιώμη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω εδώ να αναφερθώ στις συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την ιστορία αυτή, για τον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών. Όπως γνωρίζετε, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η ΛΥΜΠΕ χρειάστηκε να ασχοληθεί με πάρα πολλά νομικά ζητήματα που είχαν να κάνουν με το άσυλο και άλλα. Είναι ίσως αυτή μία εξήγηση βέβαια που οδήγησε σε καθυστερήσεις αλλά επηρέασε και τη μέθοδο και το περιεχόμενο. Υπενθυμίζω ότι στη Λίμπε είχαμε καταλήξει τον Ιούλιο του 2016 σε μια θέση και οι συζητήσεις, όπως είπατε και εσείς πρόεδρε με το Συμβούλιο, ξεκίνησαν τότε υπό τη μορφή μιας μερικής εντολής που αποκλούς, απο, απέκλειε τα μέρη των 7 χωρών που θεωρώνταν εξαρτάζονταν σαν χώρα. χώροι. Αλβανία, Ζεβοσνία, Ζεγοβίνη, Δυτικά Βαλκάνια, Μακεδονία, Κωσυβοπέδιο, ε, Μαυροβούνη, Σερβία και Τουρκία. Και όλα αυτά προκειμένου να ακούσουμε περισσότερα από τις υπηρεσίες ασύλου των χωρών αυτών. Δεχτήκαμε λοιπόν αυτήν την αρχιτεκτονική καταρχήν και θελήσαμε να δουλέψουμε βάσει τεσσάρων αρχών. Πρώτα απ' όλα τη σχέση των εθνικών καταλόγων και του ευρωπαϊκού καταλόγου, την μεθοδολογία προκειμένου να καταλήξουμε ότι μια χώρα είναι μια χώρα προέλευσης ασφαλής, τον μηχανισμό αναστολής και αλλαγή του καταλόγου εφόσον υπάρξει επιδείνωση της κατάστασης σε μια χώρα που θεωρούμε ασφαλή και τέλος το θέμα ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων των διαφερόμενων μερών. Τρεις ε, συναντήσεις είχαμε οι σκιώδεις συζητητές και οι συζητήσεις και στο τριμερή διάλογο προχωρούσαν ε, ε, καλά για το πώς καθορίζεται μια χώρα ως ασφαλής ή όχι. Προχωρήσαμε επίσης και όσον αφορά τον μηχανισμό αναστολής. Πότε δηλαδή πάβει να ισχύει ο κατάλογος αυτός ασφαλών χώρων, πότε βγαίνει ε, προσωρινά από τον κατάλογο αυτό μια χώρα. Από την άλλη, πήγαμε σημειωτών για τα θέματα της εναρμόνισης και τα θεμελιωδή δικαιώματα. Γιατί αντίθετα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντίθετα από τη δικιά του θέση, το Συμβούλιο ήθελε και θέλει πάντα νομίζω να διατηρήσει τη συνύπαρξη εθνικών καταλόγων και ευρωπαϊκού καταλόγου. Με τον κίνδυνο μάλιστα να μην λυθεί υπόψη ότι σε μερικές χώρες δεν υπάρχει καν τέτοιος κατάλογος. Και δεν προχωρήσαμε και περισσότερο ούτε για τα θεμελιώδη δικαιώματα, και το Συμβούλιο δεν θέλει να ασχοληθεί με το διαδικαστικό στα πλαίσια της υπόθεσης αυτής, αλλά θέλει να το εξετάσει στα πλαίσια του κανονισμού για τη διαδικασία. Εγώ και οι Σκιώδης, που ήταν μαζί μου και τους ευχαριστώ για το έργο τους. Για μας λοιπόν δεν μπορούσαμε να δούμε πώς είναι δυνατόν να έχουμε έναν ενωσιακό κατάλογο, χωρίς όμως να μιλήσουμε για τις διαδικαστικές συνέπειες που θα επηρέαζαν τους ανθρώπους με καταγωγή από τις χώρες αυτές. Το έχω πει και το έχουν ακούσει και συνάδελφοι που είναι σκιώδεις ε, αλλού. Το θέμα αυτό των ασφαλών χωρών γίνεται κάτι που είναι υποχρεωτικό για όλες τις χώρες μέλη, ενώ μέχρι τώρα ήταν προαιρετικό. Στη Λίμπη λοιπόν εγκρίναμε μια ισορροπημένη θέση τον Ιούλιο του 2016, λέω ισορροπημένη γιατί υπήρχε το σύστημα από τη μία και η προστασία από την άλλη των ετούντων. Και θελήσαμε όντω να υπάρχει αναρμόνιση για να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Πολύ γρήγορα από τον Νοέμβριο του 2016 καταλάβαμε ότι θα είναι δύσκολες οι συζητήσεις. Είχαμε και τη δημοσίευση της έκθεσης των γραφείων ασύλου. Και και τις μελετήσαμε αυτές τις εκθέσεις και τις αξιολογήσαμε. Χωρίς αξιολόγηση δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Οι εκθέσεις αυτές λοιπόν ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για το έργο μας και πλήρης. Επί του περιεχομένου, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις διαπιστώσεις τους ότι μία από αυτές τις χώρες, η Τουρκία, αντιμετωπίσετε προβληματικά. Τώρα, αν θέλουμε ρεαλιστικά να καταλήξουμε σε συμφωνία, εδώ αυτό φάνηκε όλο και πιο δύσκολο ο περνούσε ο χρόνος. Και δεν πρέπει όμως απ' την άλλη να αφήσουν να τρενάρουν συζητήσεις που θα αποδυνάμωναν την ε, δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη δύναμη και την όθηση με την οποία ξεκίνησε στην αρχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θέλουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας με τους σκιώδεις συζητητές, αναγνωρίζοντας ότι δεν θα πετύχουμε πρόοδο και ότι τα διέξοδα θα παραμείνουν. Η Προεδρία λοιπόν αρχέ του Μαρτίου του 2017 μα είπε, είπε ότι οι χώρε μέλη δεν θέλουν να διαπραγματευτούν άλλο και θέλουν να αναβληθεί αυτό το θέμα και να συζητηθεί στα πλαίσια του κανονισμού διαδικασία. Η Προεδρία επίσης μας είπε ότι αν οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούσαν ούτε στα πλαίσια του κανονισμού διαδικασίας, τότε θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στη θέσπιση του νοσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών. Θα δούμε δηλαδή τότε. Και για να ολοκληρώσω. Γιατί φυσικά και μας απογοητεύει το γεγονός ότι δεν μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Συγχρόνως όμως πρέπει κατά προτεραιότητα να διασφαλίσουμε ότι η θέση της ΛΥΜΠΕ γίνεται σεβαστή. Είχαμε ξεκάθαρη ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Τώρα λοιπόν πρέπει να δείξουμε ποια είναι τα δικά μας δυνατά σημεία. Το έγγραφο αυτό εργασία να το βάλουμε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το κάναμε για να μπορούν να το δουν όλοι. Και τη θέση του κ. Φεράρα νομίζω ότι με τους σκιώδες εισηγητές αποτελεί μία χρήσιμη βάση διαπραγματεύσεων για αυτό το θέμα των ασφαλών χωρών καταγωγής με την κυρία Φεράρα. Θα συνεργαστούμε πολύ επικοδομητικά πιστεύω τους επόμενους μήνες. Και τέλος ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις που με βοήθησαν και τους βοηθούς βέβαια από την πολιτική μου ομάδα που με βοήθησαν τόσο πολύ με το έργο τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω, να τώρα ε, το λόγο στην Άννα από ε, την Μαλτέζικη Προεδρία. Ε, σας ευχαριστώ πολύ ε, Πρόεδρε αλλά και την εισηγήτρια για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκφράσω τις απόψεις της Προεδρίας πάνω στο ζήτημα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και να εκφράσω την εκτίμησή μου, την εισηγήτρια, για την αποφασιστικότητα με την οποία προσεγγίσουν το συγκεκριμένο θέμα. Παρόλο, παρόλο στις προσταβάθειες όμως, ε, ο τριμερής διάλογος ε, ε, έφτασε, δεν μπόρεσε να καταλήξει παρά τις προτάσεις τον Ιούλιο του 2016. Συζητήσαμε τις ασφαλείς χώρες προέλευσης στο πλαίσιο της, υπάρχουσας, της παρούσας οδηγίας για το άσυλο. φέτος όπως ε, εξήγησε η συγγήτρια, με προσέγγισε ε, για να μου εξηγήσει ότι θα ήθελε να γίνει ένας ε, τελευταίος τριμερής διάλογος με το Συμβούλιο για να καταλήξουμε σε συμφωνία η μεθοδολογία αλλά και οι μηχανισμοί αποκλεισμού. Ενώ υπόλοιπα ζητήματα θα γινόταν στο πλαίσιο του κανονισμού για τη διαδικασία ασύλου συζητήσαμε και παρουσιάστηκε η πρόταση της γνωμοδότριας και ύστερα από μια περίοδο ε, σκέψης και συζήτησης καταλάβαμε ότι θα ήταν καλύτερο να συνεχίσουμε τη συζήτηση σχετικά με τις ασφαλείς χώρες προέλευσης ε, στο πλαίσιο του κανονισμού για το άσυλο, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους νομοθέτες να συζητήσουν τις ασφαλείς χώρες προέλευσης ε, στο πλαίσιο αυτό, αλλά και την γενικότερη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, με αποτέλεσμα να έχουμε την απαρότητη συνοχή. Έτσι λοιπόν ε, είπαμε στην γνωμοδότρια όπως ε, δηλώθηκε αλλά ε, και προς την κυρία Φεράρα στο πλαίσιο της δικής της γνωμοθέτησης ότι δόθηκε εντολή για να περιοριστούν οι, συγκεκριμέ... συζητήσεις για το συγκεκριμένο φάκελο και θα συζητηθούν ε, τα ζητήματα για τις ασφαλείς ε, χώρες ε, στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Επίσης θα θέλαμε να συζητήσουμε εάν θεωρείται αυτό αναγκαίο. Λάβαμε υπόψη μας τη θέση της γνωμοδότριας και θα το μεταφέρω αυτό και στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν έχουμε ε, ε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Ματσάρα. Αντικαθιστώ ε, την Ρωσίδα Ντάτη, ε, τη σκιώδη μας, για να σας μεταφέρω τα σχόλια όσον αφορά τη διαδικασία αυτή. Ε, κατά βάση ε, ο κοινό κατάλογος είναι ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την μεταναστευτική πίεση που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ε, δημιουργία ενό τέτοιου καταλόγου και ε, λυπούμαστε για το γεγονό ότι δεν, μπορούσαμε, δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ευελπιστούμε ότι οι συνάδελφοί μας στο EPR θα έχουν, μια καλύτερο, θα έχουν καλύτερο αποτέλεσμα στις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις. Παρ' όλα αυτά θα θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η ασυνήθιστη διαδικασία γύρει ερωτήματα, διότι ακόμα αναρωτιόμαστε πόσο συγκεκριμένος κατάλογος θα καταρτιστεί στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο ακόμα και ως σκιώδης ε, του ΕΛΚ ε, για, την, ε, για τον κατάλογο ασφαλών καταλόγων θέλουμε να δηλώσουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου και είμαστε ανοιχτοί σε διαλόγους με όλους τους συναδέλφους που εργάζονται πάνω σε, σε αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Κιέμκε. Ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση και τις προτάσεις ε, της ε, Σιλβή. Αναρωτιέμαι, μάλιστα, αν μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το κανονισμό χωρίς να συζητήσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι τόσο σημαντικό που δεν μπορούμε να κλείσουμε ένα τόσο σημαντικό φάκελο χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε με σωστά τα κριτήρια, αλλά και να συζητήσουμε και για τις χώρες ε, που έχουν ε, κατανομαστεί. Κάποιες από τις χώρες, ε, όπως η Τουρκία, η οποία συνεχώς παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία συνεχώς παραβιάζει και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, να μπει σε έναν κατάλογο ασφαλών χωρών Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Εγώ υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση της συναδέλφου. Ελπίζω ειλικρινά ότι στα πλαίσια της συζήτησης για την οδηγία να μπορούμε να κάνουμε κάποια βήματα προς τα μπρος. Αλλά αναρωτιέμαι μήπως πρέπει να θέτουμε ως κεντρικό ζήτημα το ζήτημα του σεβασμού του ατόμου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από την ε, Κομισιόν ε, αν θα θέλανε να σχολιάσουν κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μια ε, σύντομη ε, παρέμβαση. Εμείς ε, διατηρούμε την πρόταση, οπότε επαφίεται στον συνομοθέτη σχετικά με το πώς θα συνεχίσει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Okay, Ωραία, η κυρία Αρμπιόλ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κατάλογος των σίγουρων χωρών, των ασφαλών χωρών, είναι πολύ βασικό στοιχείο του μοντέλου ασύλου και μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ολόκληρο κατάλογο χωρών, ασφαλών χωρών, αλλά έχουμε παραδείγματα για το πώς έχουν συμπεριφερθεί μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Έχουμε το παράδειγμα της Τουρκίας, μια χώρα η οποία θεωρήθηκε ασφαλής, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά, τα κορίτσια που βρίσκονται εκεί ως πρόσφυγες δουλεύουν από τα 10 σε ροστάσια φαντουργίας. Αφγανιστάν. Έχουμε συμφωνία για να στέλνουμε εκεί τους πρόσφυγες γιατί θεωρούμε ότι είναι ασφαλής χώρα. Παρ' όλα αυτά η χώρα αυτή υποβάλλεται στην βία από το 2001 που πήγαν εκεί τα στρατεύματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν χρησιμοποιεί αυτό το κατάλογο για να μην έχουμε εμεί την ευθύνη να υποδεχτούμε τους πρόσφυγες, ενώ είναι δικιά μας υποχρέωση βάση του διεθνούς δικαίου. Και είναι και μία αρχή που θα χρησιμεύσει για να στρεβλώσουμε και τα θέματα του ασύλου, που είναι ατομικό δικαίωμα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχει να κάνει το αν θα δώσουμε το άσυλο ή όχι με το την εθνικότητα που έρχεται κανείς και έχει με το αν πραγματικά χρειάζεται προστασία ή όχι, όπως λέει η Σύμβαση της Γενέβης. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι είμαστε σαφώς κατά της ίδιας της αρχής αυτής των ασφαλών χωρών. Είμαστε κατά του να υπάρξει ένας τέτοιος ενωσιακός κατάλογος ασφαλών χωρών, γιατί πιστεύουμε ότι αντιβαίνει στις διεθνείς μας υποχρεώσεις και στην Σύμβαση της Γενέβης. Thank you. Uh, I would like to... Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να συζητήσω από την εισηγήτρια αν θα ήθελα να κάνει κάποια τελικά σχόλια. Ναι, ευχαριστώ, αλλά θα κλείσω πολύ γρήγορα με τρεις λέξεις. Η πρώτη, λάθος. Σε όλους τους φακέλους θα πρέπει να αποφύγουμε όλα τα λάθη, τα ενιολογικά λάθη και τα στρατηγικά λάθη. Και πιστεύω χωρίς να πάμε πιο μακριά στις εξηγήσει, ότι έγιναν κάποια στρατηγικά λάθη σε ό,τι φορά τις έννοιες σε αυτούς τους φακέλους. Το δεύτερο είναι η παναχώρηση. Το να επαναχωρήσουμε σε αυτούς τους φακέλους δεν θα αλλάξει τίποτα, δεν θα μας επιτρέψει την επίλυση των θεμάτων αυτών, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Και το τρίτο είναι αποφασιστικότητα. Ό,τι και να γίνει, Πιστεύω ότι η ομάδα συζήτηση ε, για το νομοθέτημα για τις διαδικασίες ασύλου ε, ουσιαστικά πρέπει να ληφθεί υπόψη και φυσικά πρέπει να δούμε τι έχουμε κάνει και εκεί σε σχέση με τον ορισμό των ασφαλών τρίτων χωρών. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τώρα να περάσουμε στο σημείο 16. Έχουμε 15 λεπτά στη διάθεσή μας. Στις 5 Ιουλίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για μια απόφαση του Συμβουλίου για το Πολιετές ε, Πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022. Αυτό το Πολιετές ε, Πλαίσιο θετείται κάθε πέντε χρόνια και ορίζει τους θεματικούς τομείς ε, της δραστηριότητας του οργανισμού. Στις 28 Νοεμβρίου υιοθέτησε το Συμβούλιο το σχέδιο απόφασης, ε, το οποίο, η οποία θα υιοθετηθεί οριστικά δυνάμει του άρθρου 352. Η Προεδρία του Συμβουλίου παρουσίασε το σχέδιο απόφασης στη συνάντησή μας στις 31 Ιανουαρίου και σήμερα η κυρία Μιλάρ θα παρουσιάσει το σχέδιο της γνωμοδότησής της. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν, ε, θέλω να ευχαριστήσω την Προεδρία της ε, Μάλτας για την ε, δέσμευσή της, την Κομισιόν για τη συνεργασία της και τους κοιότητες για την υποστήριξη όπως έχει αναφερθεί σε άλλες περιπτώσεις. Εγώ λυπάμαι για την έλλειψη συμφωνίας στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη των θεματικών της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές αποθέσεις στο νέο πολιετές πλαίσιο. Η συμπερίληψη της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας στο πολιετές πλαίσιο όχι μόνο θα αντικατόπτριζε τι τις ανάγκες επιτόπου, αλλά και θα επέτρεπε στον οργανισμό να δώσει πλήρες αναλύσεις σε τομείς που είναι φυσικά πάρα πολύ σχετικοί με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, θα έστελνε και το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τις πτυχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία και σε ποινικά ζητήματα. Σίγουρα αυτό το επιθυμούν και το αναμένουν και οι πολίτες αλλά η κοινότητα των ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάντως, εν απουσία ενός ε, νέου πολιετούς πλαισίου στις αρχές του 2018, ο οργανισμός θα μπορούσε να εργαστεί μόνο επειδή υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα από κάποιο οργανισμό και όχι δύο πρωτοβουλία. Και φυσικά αυτό δεν μας συμφέρει και θα πρέπει να αποφευχθεί. Προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτό το μηχανισμό χωρίς να υποσκάψουμε το έργο του οργανισμού. Εγώ ξεκίνησα έναν επικοδομητικό διάλογο με Συμβούλιο και Κομισιόν και καταλήξαμε σε μια συμφωνία καθώς και τα δύο όργανα θέλουν να δεσμευτούν για την ε, τροποποίηση του ιδρυτικού μηχανισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για να αντικατασταθεί η αναφορά στην ευρωπαϊκή κοινότητα και να δημιουργηθεί μια, ένας οργανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή ε, και να περιλαμβάνονται και θέματα αστυνομικής συνεργασίας, ε, πρώην τρίτου πυλώνα δηλαδή, και να βελτιωθούν οι διαδικασίες για την λειτουργία του οργανισμού έχει ζητηθεί να υπάρξει μία δήλωση ε, και να διαβαστεί η δήλωση εδώ σήμερα στην Επιτροπή. Θέλω να ενημερώσω τους Κιώδης και να ζητήσω να έχουμε μία δήλωση Συμβουλίου και Κομισιόν ε, στην Μήνυ Ολομέλεια του Μαΐου. Αυτό θα μας επιτρέψει ε, ως Κοινοβούλιο να τοποθετηθούμε και εμείς μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, θέλω να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Κομισιόν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Θέλω να κάνω την ακόλουθη δήλωση εκ μέρους της Κομισιόν. Η Κομισιόν λυπάται την έλλειψη συμφωνίας για τη συμπερίληψη της προτινόμενης ε, νέας θεματικής της αστυνομικής συνεργασίας και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στο πολιτέ πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2018-2022. Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι Κατόπιν τη θέσεω ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνη, η αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει έχει καταστεί μέρο του ενωσιακού δικαίου και επομένω καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογή των καθηκόντων ε, του οργανισμού δυνάμει του άρθρου 3.1 του κανονισμού 168-2007. Αν αυτοί οι θεματικοί τομεί δεν συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση του Συμβουλίου που θεσπίζει το πολιετέ πλαίσιο για τον οργανισμό για την περιοδο 2008 2018-2022, ο οργανισμός θα συνεχίσει να υλοποιεί τα καθήκοντά του σε αυτούς τους τομείς κατόπιν αιτήματο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, ή την Κομισιόν, δυνάμει του άρθρου 53 του ίδιου κανονισμού. Όμως, κατόπιν εξωτερικής αξιολόγησης του οργανισμού το 2017, η Κομισιόν θα στείλει και τις εκθέσεις αξιολόγησης και τις συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο, στην ΕΟΚΕ και στην Επιτροπή των Περιφερειών και θα τα δημοσιεύσει τα εγγραφά αυτά. Κατόπιν της αξιολόγησης, της έκθεσης αξιολόγησης και των συστάσεων, η Κομισιόν ίσως να στείλει προτάσεις τροποποίησης του κανονισμού 168-2007, αν το θεωρήσει απαραίτητο, έτσι όπως προβλέπεται στο άρθρο 312. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Κατρίνα Μιζικρήμα από την Μαλτεζική Προεδρία. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους τη Προεδρίας ε, θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο, καθώ και την εισηγήτρια. Δυνάμει του άρθρου 30, παράγραφη 3 και 4 του κανονισμού του Συμβουλίου 168, καθ 2007, ο κανονισμό προτείνει ότι γίνεται μία αξιολόγηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στο 31 παράγραφος 2. Η Κομισιόν, αφού θα έχει κάνει εξέταση της έκθεσης αξιολόγησης και της συστάσεις, μπορεί σε αυτή τη βάση να υποβάλει προτάσεις τροποποίησης του κανονισμού, τις προτάσεις που θεωρεί απαραίτητες. Στα πλαίσιο αυτό αυτό το Συμβούλιο θα εξετάσει οποιασδήποτε προτάσει τροποποίησης του κοινωνισμού που μπορεί να στείλει Κομισιόν και ε, σε ό,τι αφορά την κάλυψη των τομέων της αστυνομικής δικαστικής συνεργασίας σε ποινικέ υποθέσεις. Το Συμβούλιο θα εξετάσει προσεκτικά οποιασδήποτε προτάσεις για τη βελτίωση της ε, λειτουργίας ε, και της διαχείρισης του οργανισμού, της δίκησης του οργανισμού. Ωραία, ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στη συζήτηση. Η κυρία Μετσόλα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Βάρβαρα. Εγώ αντικαταστώ τον κύριο Νάτζη. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ε, δουλειά σας, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, ουσιαστικά προσφέρει πολλά στα θεσμικά όργανα, η έρευνά του και η δουλειά του και η παροχή συμβουλών σε συγκεκριμένους τομείς υποστηρίζουν την καθημερινή δουλειά μας. Ο κύριος Νάτς θεωρεί ότι προς στιγμή δεν υπάρχει νομική βάση τροποποίησης ή να προσθέσουμε περαιτέρω ε, αρμοδιότητες ε, στο ΦΡΑ μέσω του πολιτού πλαισίου, όμως υποστηρίζει πλήρως την εισηγήτρια και θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση εάν υπάρξει βούληση μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Thank you for such concrete statement. Ευχαριστώ για τη δήλωσή σας, ε, η κυρία ε, Σούπα. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς η ε, δική μας σκιώδης δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας και γι' αυτό το λόγο θα μιλήσω εκ μέρους της. Θα ήρθε αρχικά να, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια αφενός για το ότι έγραψε το προσχέδιο ε, και ε, για το γεγονός ότι έλαβε υπόψη της ε, τον ιδιαίτερο ρατσισμό που απευθύνεται στους Ρωμά και την περιθωριοποίηση που αντιμετωπίζουν και που το περιλαμβάνει αυτό στην ε, θεματική ε, για την ε, ενσωμάτωση των ΟΜΑ. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Μίλνερ για την ώρα για το ότι άσκησε ποιήση τόσο στην Κομισιόν όσο και στο Συμβούλιο για να υπογράψουν μια κοινή διακήρυξη η οποία εγκρίνει την συγκεκριμένη συνθήκη για, τα, για τον τρίτο πυλώνα. Θα πρέπει να συμπληρωθούν αυτά τόσο στην αστυνομική όσο και στην δικαστική συνεργασία. Ε, τώρα με βάση όλων αυτών η ομάδα μας θα υποστηρίζει την πρόσταση της εισηγήτριας ε, να ε, εγκριθεί η απόφαση του Συμβουλίου σε περίπτωση που τόσο ε, η Κομισιόν όσο και το Συμβούλιο τηρήσουν την υπόσχεσή τους. Ευχαριστώ. Ναι, και ο κύριος Κρύπακ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν πάνω σε αυτό το φάκελο ε, και εκφράζουμε την ε, ε, υποστήριξη του ECR για την θέση αυτή και για το ότι δεν θα πρέπει να αυξηθεί η εντολή. Επίσης θα πρέπει θεωρούμε ότι ο κανονισμός είναι αποτελεσματικός και αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε τη συγκεκριμένη πεποίθηση. Ε, η νομοδότρια έχει συμφωνήσει ε, να συνεργαστεί με την υπηρεσία, όμως ε, θεωρούμε ότι ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να επεκταθεί, να αλλάξει. Δεν θα υποστηρίξουμε αυτό το κομμάτι του προσχεδίου και θα υποβάλουμε τις αντίστοιχες τροπολογίες. Η κυρία Λούνατσεκ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Χνομοδίτρια για την προσέγγιση της ε, θέλοντας να ασκήσει πίεση στο Συμβούλιο για να περιλάβει όπως ε, θεωρούμε εμείς ε, και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικά ζητήματα για πολλούς εξημών το σωστό να γίνει. Όμως πριν κάνω αυτό θα ήθελα ε, να ε, υποστηρίξω ιδιαίτερος ε, την υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα η οποία παρέσχει σημαντικό έργο και για τη δουλειά που κάνουμε εμείς παρόλο που υπάρχουν μερικοί οι οποίοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να το αγνοήσουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Παράσχουν πολύ σημαντικές έρευνες ε, για τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα ε, για πάρα πολλές ε, ομάδες, για όλες τις ομάδες που βιώνουν διακρίσεις αυτή την Ήπειρο τόσο για τα κράτη-μέλη, ε, είτε ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μιλάμε για ε, μέλη της κοινότητας ΛΟΑΔΜΑ, για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, για τους Ρωμά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας είτε στη ΛΥΜΠΕ, είτε σε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή χωρίς το έργο της υπηρεσίας και γι' αυτό το λόγο εκτιμώ τα όσα λέει η ε, έκθεση το ότι χρειαζόμαστε τη συγκεκριμένη υπηρεσία ε, και ως πράσινοι αλλά και άλλες ομάδες ε, θα θέλαμε η εντολή της υπηρεσίας να είναι ακόμα πιο ισχυρή. Ας αγωνιστούμε για αυτό. Ε, όπως και να έχει εγκρίνουμε επίσης ε, τα όσα μας ζήτησε η συγγήτρια, ε, δηλαδή να υποστηρίξουμε το κείμενο και τα όσα είπε το Συμβούλιο, να εξετάσουμε δηλαδή, με το, να εξετάσουμε τρόπους με τους οποίους το Συμβούλιο μπορεί να κινηθεί προς τα εμπρός και να έχουμε και το ζήτημα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας ε, δεν μετανιώνω το πώς είναι τώρα, όμως ε, εμείς ως ομάδα το εγκρίνουμε. Ευχαριστούμε και η κυρία Σπινέλη τώρα. Ευχαριστώ την κυρία Μλίναρ για το θεραλέο έργο της και υποστηρίζω πλήρως τις συστάσεις που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, στο σχέδιο έκθεσης. Δύο σημεία είναι πάρα πολύ σημαντικά και για μένα όπως και για την συγκέντρια. Καταρχήν, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μεταξύ των συστηματικών τους ε, του πολιετούς πλαισίου να μπορεί να συμπεριλαμβάνει το θέμα της κοινωνικής ε, ένταξης ε, των Ρωμά και να υποστηρίξει ΟΦΡΑ, το κέντρο κατά της αθηκανοφοβίας για να μπορέσουν να καταπολεμηθούν οι αιτίες ε, ρατσισμού και περιθωρήσεις των Ρωμά. Δεύτερο, Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε στο νέο πολιετές πλαίσιο τους θεματικούς τομείς της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας ε, και όχι μόνο στις αστικές αλλά και στις ποινικέ υποθέσεις και αυτό θα επέτρεπε να συμπεριλάβουμε στο έργο του οργανισμού θέματα που είναι πολύ σημαντικά για την ασφάλεια της Ένωσης, κατά πολέμηση της μαφίας, της απάτης, κατά της τρομοκρατίας κτλ. Δεδομένου των τελευταίων νομοθετικών προτάσεων της Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και αν λάβω υπόψη το πόσο επηρεάζουν αυτές οι πολιτικές ε, στο θέμα της ιδιωτικότητας της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και στα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων και των ανηλίκων, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και επιβεβαιώνω πλήρως ότι η ΜΚΟ πρέπει να δώσουν μεγάλη σημασία ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να μπορεί η Δία Πρωτοβουλία να αναπτύσσει μελέτες για αυτή τη θεματική. Κλείνω λέγοντα ότι και εγώ απογοητεύτηκα από το γεγονό ότι το Συμβούλιο δεν κατέληξε σε συμφωνία για τη συμπερίληψη αυτού του τομέα στο πρόγραμμα του οργανισμού. Όμως, ε, καθώς ε, θεωρώ ότι δεν πρέπει ποτέ να ε, υποχωρούμε, εμπιστεύομαι τους εαυτούς μας ότι μπορούμε να σκίσουμε πειθό και είμαι πεπισμένη ότι η Αγγέλικα έχει την ε, ικανότητα και την αποφασιστικότητα να κάνει αυτή τη διαδικασία πειθούς. Την υποστηρίζω λοιπόν πλήρως. Σας ευχαριστώ. And the end, Mrs. Η κυρία Κέγγε. Ευχαριστώ. Και εγώ να πω ότι υποστηρίζω πλήρως ε, και έχω θετική απόκριση στα όσα υποστήριξε η δική μου ομάδα. Όμως θέλω να επενθυμίσω και στον Οργανισμό Θεμελιών Δικαιωμάτων, αλλά και σε όσου εργάζονται σε αυτό τον τομέα, ότι σήμερα έχουμε μια καλή στρατηγική καταπολέμηση του ρατσισμού. Δηλαδή, αναγνωρίζονται όλε οι μορφέ ε, εισαγωγή διακρίσεων. Είναι δύσκολο στη βιβλιογραφία να βρούμε ε, θέμα, ε, το, το θέμα του ρατσισμού κατά ανθρώπων που προέρχονται από την Αφρική. Λέγεται αφροφοβία. Έτσι λοιπόν σήμερα πρέπει να έχουμε μία πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Αυτό το λέω όχι γιατί πρέπει να επικεντρωθούμε σε μία κοινότητα, αλλά πρέπει να κατονομάσουμε όλες τις μορφές ρατσισμού και διακρίσεων. Αν αφήσουμε κάποια εκτός, η πλήρης καθολική στρατηγική δεν θα έχει νόημα. Και γι' αυτό Σήμερα εφιστώ την προσοχή σας ε, στο σημείο αυτό, το profiling αφορά κυρίως ανθρώπους με αφρικανική καταγωγή, με χαρακτηριστικά που είναι αναγνωρίσιμα και γίνονται εύκολα θύματα λόγω αυτής της δημιουργίας προφίλ. Ζητώ λοιπόν εδώ να ληφθούν υπόψη πέρα από όλες τις μορφές που παρουσιάστηκαν και η πραγματικότητα της ε, αφροφοβίας ε, που είναι παρούσα ακόμη και αν δεν συζητείτε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής ε, έχουν μια πραγματικότητα και δεν είναι δυνατόν να την κρύψουν. Ευχαριστώ. Η Αγγέλικα τώρα. Μήπως θέλετε να καταλήξετε σε συμπεράσματα ολοκληρώνοντα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, ευχαριστώ για τη στήριξη. Και ξέρετε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η αποτυχία δεν είναι επιλογή, οπότε πρέπει να πετύχουμε. Τίποτα άλλο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 20 Απριλίου 2017 στις 3 το μεσημέρι. Και σημειώστε ότι πρόκειται για τη σύμφωνη γνώμη. Οι τροπολογίες δηλαδή πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Word, στο σύστημα Word και όχι σε κανένα άλλο. Εντάξει. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλό και Πάσχα. Γεια σας. Do you know that we continue this... Αλλά ξέρετε ότι και σήμερα το απόγευμα συνεχίζουμε, έτσι.